συνάδελφοι, Καλώς ήρθατε λοιπόν και ξεκινούμε τη συνεδρίαση με την έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Θεωρούμε ότι εγκρίθηκε και σας ευχαριστώ. Καλώς ορίζω τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, κύριο Μάριο Τράγκη. Τον ευχαριστώ που είναι εδώ για το δεύτερο νομισματικό διάλογο του έτους. Όπως θα θυμάστε, ο προηγούμενος είχε λάβει χώρα στις 6 Φεβρουαρίου. Σήμερα ο σημερινό θα ακολουθηθεί και από μια δημόσια κρόση με τον κύριο Μαρίο Ντράγκη ως πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου. Όπως όλοι γνωρίζουμε από τον τελευταίο νομισματικό διάλογο έχει διατηρήσει χωρίς αλλαγές στι θέσεις της η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και σε σχέση με τα μέτρα νομισματικής πολιτικής. Το Νομισματικό Συμβούλιο ξέρουμε ότι έχει επιβεβαιώσει πως τα μέτρα αυτά θα διατηρηθούν έως το τέλος του χρόνου και ενδεχομένω να παρατεθούν, εάν καταστεί απαραίτητο. Και πάντως θα συνεχίσουν μέχρι να εξασφαλιστεί επαρκής προσαρμογή στους ρυθμούς του πληθωρισμού και, μέχρι, και βεβαίως το Συμβούλιο είναι διατεθειμένο να ε, συνεχίσει το πρόγραμμα εξαγοράς τίτλων. Είναι λοιπόν μέτρια αλλά σταθερή αυτή η ανάκαμψη της Ευρωζώνης, δεν πρέπει να τεθεί σε κίνδυνο. Υπάρχουν επαρκή μέσα για την αντιμετώπιση κάθε πολιτικής ή γεωπολιτικής έκτακτης ανάγκης. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με τις μη συμβατικές της πολιτικές έχει δραματίσει κρίσιμο ρόλο στην υποστήριξη της ιστορικής ζήτησης και ουσιαστικά έχει βοηθήσει στην μόχλευση στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα της οικονομίας, μια πολιτική η οποία θα πρέπει να οδηγήσει σε επίπεδα αντίστοιχα με τους στόχους της ΕΚΤ. Θα μας παρουσιάσει ο κύριος Τράγκη λοιπόν τους, ε, την προοπτική προς τις οικονομικές και νομισματικές εξελίξεις, θα σχολιάσει τις συνέπειες του Brexit για την ε, σταθερότητα τη χρηματοπιστωτική της ε, Ευρωζώνης. Επίσης θα επεκταθεί και σε θέματα που έχει επιλέξει η Επιτροπή μας εν ώψη αυτού του νομισματικού διαλόγου, δηλαδή την χρηματοπιστωτική καινοτομία και τις συνέπειες για την νοσματική πολιτική και το ζήτημα εάν η αύξηση των μακροπρόθεσμων ε, επιτοκίων είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα ή αντίξωμα αποτελέσματα. Έχουμε σημειώσει ότι η παρατηρούμενη αύξηση των μακροπρόθεσμων επιτοκίων από τον Αύγουστο του 2016 παρατηρείται αποδίδεται και στην αύξηση των αντίστοιχων επιτοκίων των πολιτικών μετά την αλλαγή της νομισματικής τάσης της ΦΕΔ, αλλά ταυτόχρονα οφείλονται και σε πολιτικές εντάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θεωρούνται ως υψηλός πολιτικός κίνδυνος και μπορεί να παραμένουν αυτά τα στοιχεία, αλλά μπορεί ο πολιτικός κίνδυνος με τις προσεχείς εκλογές αλλά και τις την τελευταία εκλογική αναμέτρηση να υποχωρήσει. Υπογραμμίζεται επίσης η ιδέα ότι το να σταματήσει πρόωρα το QE, η ε, οικονομική διευκόλυνση, μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις. Έχουμε πολλά ενδιαφέροντα θέματα λοιπόν και η ποσοτική χαλάρωση. Και βεβαίως περιμένουμε τώρα από τον ε, κύριο Δράκη να μας κάνει την παρουσίασή του. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Πρόεδρε, αγαπητοί κυρίε και κύριοι, μέλη τη Επιτροπή ε, των Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων, κυρίε και κύριοι, με χαρά έρχομαι να σα ξαναμιλήσω ω ε, πρόεδρο του ε, Συμβουλίου Ευρωπαϊκού Συντομικού Κινδύνου για αυτό το δεύτερο διάλογο. Χαίρομαι ιδιαίτερω που έχετε επιλέξει ω τίτλο τον ρόλο της ε, οικονομικής καινοτομία, τη οικονομική καινοτομία Πρόκειται για έναν από του ρόλου καινοτομία που μπορεί να στηρίξουν την οικονομία, πρόκειται για έναν αποφασιστικό ρόλο δεδομένου του αισιόδους ρόλου των χρηματοπιστωτικών αγορών ω προς την κατανομή των πόρων. Πριν να επεκταθώ στο θέμα αυτό, επιτρέψτε μου πρώτα να αναφερθώ στις οικονομικές προοπτικές και να ε, τοποθετηθώ ως προς την ε, οικονομική πολιτική. Η ανάκαμψη ενδυναμώνεται και διευρύνεται σε τομείς και χώρες. Το πραγματικό ΑΕΠ στην Ευρωζώνη επεκτείνεται επί 16 συνεχόμενα τρίμηνα, 1,7% ανάπτυξη κάθε χρόνο, κατά το, και κατά το πρώτο τρίμηνο του 2017. Η ενεργεία έχει πέσει στο χαμηλότερο από το 2009 επίπεδο. Η εμπιστοσύνη των καταναλωτών και των επιχειρήσεων έχει αυξηθεί, έχει φτάσει σε επίπεδο υψηλότερο των 6 τελευταίων ετών και αυτό υποστηρίζει την ιδέα μιας περαιτέρω ενίσχυσης ανάπτυξης για τους επόμενους μήνες. μειώνονται οι κίνδυνοι και η πολυματική κίνδυνη που είχαμε αντιληφθεί στο τέλος του προηγουμένου έτους φαίνεται να είναι συγκρατημένη. Το γεγονό ότι η εσωτερική κατανάλωση και οι επενδύσεις αποτελούν τους κύριους κινητήρες της ανάπτυξης την καθιστούν πιο ε, στεναρή, πιο ανθεκτική στους εξωτερικούς κινδύνους που βέβαια συνδέονται κυρίως με παγκόσμιους ε, παράγοντες και στοιχεία. Παρά την περαιτέρω ανάκαμψη λοιπόν και με την πτυτικότητα που διαπιστώνουμε, ιδιαίτερα στον ε, πληθωρισμό, πρέπει να πούμε ότι ο πληθωρισμός έχει παραμείνει συγκρατημένος. Η εσωτερική πίεση στο κόστος, κυρίως από τους μισθούς, είναι ανεπαρκής και δεν μπορεί ακόμη να στηρίξει ε, βιώσιμη και αυτό ε, ανάπτυξη προς τους νοσοπρόθεσμους στόχους μας σε σχέση με τις πιέσεις τώρα το, στις τιμές. Για να ενισχυθούν αυτές χρειάζονται πιο κατάλληλες οικονομικές συνθήκες που εξαρτώνται οι ίδιες από, ουσιαστικό, ε, από ουσιαστική και παρακολούθηση της νομισματικής πολιτικής. Το Διοικητικό Συμβούλιο λοιπόν λαμβάνει και επικαιροποιεί τις προβολές που υποβάλλουν το προσωπικό του σε ένα σύστημα, σε ένα ε, σύνολο που του επιτρέπει να κατανέμει, να εξετάσει καλύτερα την κατανομή του κινδύνου πέραν της ε, ανάκαμψης και των κινδύνων από τον πληθωρισμό. Παραμένουμε πεπισμένοι ότι η υποστήριξη με την νομισματική πολιτική βέβαια και με τη δική μας καθοδήγηση θα χρειαστεί να συνεχιστεί δεδομένης ε, της ε, μη απορρόφησης των πόρων αυτή τη στιγμή και για να μπορέσει ο πληθωρισμός να γυρίσει σε επίπεδα σταθεροποιημένα γύρω στο 2% μεσοπρόθεσμα. πρόθεσμα. Μου ζητήσατε σήμερα να σας παρουσιάσω τη δυναμική των μακροπρόθεσμων επιτοκίων. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες η απόδοση των μακροπρόθεσμων ομολόγων είχε επιτοτική τάση και σε ονομαστική αλλά και σε, ονομαστικούς αλλά και σε πραγματικούς όρους. Και ενώ η χαμηλότερη απόδοση αντικατοπτρίζει την εμπορική βέβαια πολιτική, η υποχώρηση τα τελευταία χρόνια καθοδηγείται από διαρθρωτικούς παράγοντες, οι οποίοι έχουν να κάνουν και με την αύξηση των καθαρών ε, αποθεμάτων αποταμίευσης, καθώς ε, γυράζει και ο πληθυσμός, και ε, τον περιορισμό στις κρατικές δαπάνες λόγω του χρέους, αλλά και την υποχώρηση της ανάπτυξης. Για να αυξηθούν λοιπόν και πάλι τα επιτόκια σε βιώσιμα επίπεδα, πρέπει να αντιμετωπιστούν οι λόγοι των προβλημάτων και αυτό σημαίνει διαθροτική δράση σε εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η νομισματική μας πολιτική από πλευρά της είχε κρίσιμο ρόλο στην αντιμετώπιση του κυκλικού συστατικού τη στάθμιση μεταξύ της εξασφάλισης ε, αποταμίευσης και των, ε, της ζήτησης και με την υποστήριξη των ονομαστικών εισοδημάτων, ε, τα μέτρα μας, νομισματικής πολιτικής μέτρα, ενισχύουν την κατανάλωση. Μία προϋπόθεση για την ανάκαμψη του πληθωρισμού σε επίπεδα χαμηλότερα μεν, αλλά κοντά στο 2%. Μια πιο δυναμική πολιτική, οικονομία δηλαδή, θα έχει καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με τα επιτόκια. Τώρα θα ήθελα να περάσω στην σημασία της οικονομικής καινοτομίας. Η σχέση μεταξύ αποταμίευσης και επενδύσεων με οδηγεί στο θέμα το οποίο επιλέξατε για τη σημερινή σας ακρόαση και η αποτελεσματικότητα της χρηματοπιστωτικής λειτουργίας στην Ευρωζώνη σημαίνει και ε, παραγωγή κεφαλαίου και χρήση του κεφαλαίου αυτού κατά τρόπο παραγωγικό η καινοτομία στα χρηματοπιστωτικά μέσα, τις υπηρεσίες, τις υποδομές, αλλά και οι αλλαγές στην οργάνωση των χρηματοπιστωτικών ε, αγορών ε, μπορεί να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο, χρήσιμο ρόλο. Στην περίπτωση αυτή η χρηματοοικονομική καινοτομία είναι μια συνεχιζόμενη διαδικασία. Έχει στο παρελθόν πάντοτε ακολουθήσει ενωδικές στάσεις και είχαμε παραδείγματι την εισαγωγή των διασφαλιζόμενων χρεών, των ε, ε, μετοχών με προτίμηση που προσελκύουν περισσότερο τους ενδιαφερομένους και αντικσταθμίζουν τις ασυμμετρικές τάσεις. Άλλες καινοτομίες έχουν μειώσει το κόστος των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και έχουν καθιταστεί κομμάτι της καθημερινής μας ζωής. Πιστωτικές κάρτες, Φιλιππίν, ή ATM, μηχανήματα ανάληψης. Τώρα με την καινοτομία και τη νέα τεχνολογία για την, που χρησιμοποιείται πλέον στις οικονομικές ε, υπηρεσίες και τις τράπεζες, μπορούμε να πούμε ότι έχουμε μία δύναμη μετατροπής. Παρακολουθούμε βεβαίως ε, τις εξελίξεις για διάφορους λόγους και για να καταλάβουμε καλύτερα τι είδους επιπτώσεις μπορεί να έχει και για να αξιολογήσουμε τους κινδύνους και για να προσαρμόσουμε το ρυθμιστικό πλαίσιο και την εποπτική προσέγγιση όπου αυτό χρειάζεται. Και ταυτόχρονα για να προσαρμόσουμε ως θεσμός και να προσαρμοστούμε ως θεσμός και να υποστηρίξουμε την καινοτομία που αυτό χρειάζεται. Μερικά συγκεκριμένα παραδείγματα λοιπόν, γιατί η FinTech έχει άμεσο αντίκτυπο στη δική μας δουλειά. Ε, μια εις βάθος γνώση του τρόπου με τον οποίο η χρηματοοικονομική πολιτική επηρεάζει την πραγματική οικονομία έχει κρίσιμη σημασία για μας. Η FinTech και γενικότερα η χρηματοοικονομική καινοτομία έχουν δυναμικό για να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο χρηματοδοτείται η πραγματική οικονομία και μπορεί να επηρεάσουν τους μηχανισμούς της οικονομικής πολιτικής και τους όρους της χρηματοδότησης τελικά. Ως ε, Κεντρική Τράπεζα λοιπόν της Ευρωζώνης διατηρούμε την ε, επαγρύπνησή μας βεβαιόμενοι ότι το οικονομικό περιβάλλον βρίσκεται υπό έλεγχο και εποπτεία. Η ΕΚΤ και το Ευρωσύστημα επίσης έχουν ε, θεσμικό ενδιαφέρον για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των συστημάτων πληρωμής και των υποδομών των αγορών. Ένα από τα πιο δραστήρια πεδία καινοτομία της FinTech που μπορεί να αφορά τις πληρωμές και τις ε, μετοχές είναι τα συστήματα για τα ουλής μετοχές TLT όπως το blockchain. Είναι ταχύς η ρυθμή ανάπτυξης και γι' αυτό πρέπει να παρακολουθούμε διαρκώς και να αξιολογούμε νέους ή και πιο έντονους ε, εντεταμένους κινδύνους όπως ε, το σύστημα TLT to payment, το clearing ε, και άλλα. Ένας κίνδυνος λοιπόν τέτοιου τύπου θα ήταν η αύξηση του κατακαιρματισμού των αγορών. Εάν εγκαθιδρυκθούν διαφορετικές προσεγγίσεις DLT σε διαφορετικά κρατημέλη. Επιπλέον, το σύστημα εποπτείας του ευρωσυστήματος πρέπει να διτηρήσει την αποτελεσματικότητά του για να μπορέσουμε να επιτελέσουμε το καθήκον μας σε αυτό το νέο περιβάλλον. Το ευρωσύστημα βεβαίως θα συνεχίσει να δρά βάσει της συντολής του για την προαγωγή της απρόσκοπτης λειτουργίας των συστημάτων πληρωμών. Επίσης η FinTech εξασφαλίζει για τον χρηματοοικονομικό τομέα γενικότερα τη δυνατότητα για πιο αποτελεσματικές, πιο αποδοτικές υπηρεσίες για τα νοικοκυριά ή τις επιχειρήσεις. Η FinTech μπορεί επί παραδείγματι να διευκολύνει μια τράπεζα στην προσαρμογή του επιχειρησιακού της μοντέλου, την περικοπή του κόστου, στην αξιοποίηση νέων επιχειρηματικών ε, ευκαιριών. Οι εταιρείε FinTech μπορούν επίσης να συμπληρώσουν ε, την δανειοδοτική δυνατότητα των τραπεζών προσφέροντας ένα νέο ε, μέσο πρόσβασης ε, στις, στη χρηματοδότηση, παραδείγματι με πλατφόρμες peer-to-peer -peer, to peer ισοτήμων για την δανειοδότηση. Και έτσι μπορεί να αντισταθμιστεί η μείωση των δυνατότητων δανειοδότηση από τις τράπεζες προς τα νοικοκυριά, περιλαμβανομένων και των μικρότερων τραπεζών. Επίσης, η όλο και μεγαλύτερη σημασία των μη τραπεζικών φορέων και η επέκτασή του σε άλλες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες μπορεί να ενέχουν και νέους κινδύνους. Έτσι λοιπόν είναι απαραίτητο να αξιολογηθεί και να προσαρμοστεί το κανονιστικό πλαίσιο προκειμένου να καταγραφεί σωστά ο αυξανόμενος ε, παράγων κινδύνου που μπορεί να ενέχουν αυτές οι μη τράπεζες, να καταγραφούν οι νέοι παράγοντες και να εξασφαλιστούν τα κατάλληλα μέτρα και μέσα για την αντιμετώπιση των νέων κινδύνων. Για το σκοπό αυτό λοιπόν συμμετέχουμε δραστήρια σε συνεχιζόμενο έργο σε επίπεδο ευρωπαϊκό αλλά και διεθνές. Πέραν αυτού, κίνδυνος που απορρέει από τη χρήση των νέων τεχνολογιών θα πρέπει να τύχει προσεκτικής διαχείρισης, ιδιαίτερα όσον αφορά τους κινδύνους που μπορεί να προέρχονται από την κυβερνο, κυβερνοασφάλεια. Η, η κυβερνοασφάλεια λοιπόν έχει πολύ μεγάλη σημασία για τις εθνικές αρχές, αρχές ιδιαίτερως υπεπτίας και από την πρώτη στιγμή η εποπτεία της ΕΚΤ έχει εξετάσει το θέμα αυτό από τις διάφορες πτυχές του ως αρχή εποπτική των υποδομών των αγορών εξετάζουμε αν ο πολίτης ως μεμονωμένο άτομο αλλά και το δίκτυο ολόκληρο έχει ε, ανθεκτικότητα επαρκή στο κυβερνοέγκλημα. Παρακολουθούμε λοιπόν τους κινδύνους που μπορεί να προκύπτουν από τη FinTech. Ταυτόχρονα όμως συμβάλλουμε και στην χρηματοοικονομική καινοτομία ως παράγοντες που συμμετέχουν σε αυτήν. Ο στόχος για την ε, πλατφόρμα TT2S ε, που ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2015 είναι ακρογωνιά ακρογωνιαίος λίθος ε, της οικονομίας της αγοράς και έχει ιδιαίτερα βοηθήσει στην προαγωγή και τη δημιουργία εναρμονισμένων, ολοκληρωμένων και αποτελεσματικών συστημάτων πληρωμών και τίτλων. Επίσης η ΕΚΤ δρά καταλυτικά στη δημιουργία μιας πραγματικής γνήσιας ευρωπαϊκής αγοράς για τις πληρωμές και τους τίτλους. Η χρηματοοικονομική λοιπόν ε, σταθερότητα, η χρηματοοικονομική αγορά είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους πολύ στενά. Πρέπει να έχουμε βέβαια κανονιστικό πλαίσιο και πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η χρηματοοικονομική ενοποίηση και ανάπτυξη ενισχύουν η μία την άλλη και έτσι βελτιώνουν την ε, αποδοτικότητα του χρηματοοικονομικού συστήματος. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο ο νομοθέτης Ευρωπαϊκής Ένωση έχει να διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο. Ένα εναρμονισμένο πλαίσιο, ένα πλαίσιο στηριζόμενο σε αρχές σε σχέση με τη FinTech, εναρμονισμένο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, μαζί με το σχετικό θεματολόγιο θα μπορέσει να εξασφαλίσει ένα πεδίο ισότιμου ανταγωνισμού εξ αρχή, πράγμα το οποίο θα ενισχύσει με τη σειρά του τις διασυνοριακές επενδύσεις και τη διασυνοριακή επέκταση της αγοράς. Όπως βλέπετε λοιπόν η FinTech έχει δυναμικό να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα στον χρηματοπιστωτικό τομέα, να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες, να μειώσει την τιμή για τον καταναλωτή, τις τιμές για τον καταναλωτή, αλλά έχει και άλλες διαστάσεις σε σχέση με τη διαμόρφωση νέων κινδύνων και την αντιμετώπιση με ρυθμιστικό τρόπο, με κανονιστικό τρόπο αυτών. Καθήκον μας είναι να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις. Όλος ο χρηματοπιστωτικός τομέας εξαρτάται από αυτόν καθώς επεκτείνεται η φύντη και θα χρειαστούν πολλαπλές και διαφορετικές ε, μορφές ανταπόκρισης και αντίδρασης. Πρέπει λοιπόν να έχουμε και προληπτική δράση, προστασία του καταναλωτή αλλά και άλλους ε, κανονισμούς και ρυθμίσεις, χωρίς ωστόσο να παρεμποδίσουμε τις εξελίξεις. Και για να καταλήξω, οι οικονομικές προοπτικές για την Ευρωζώνη είναι θετικές, είναι περιορισμένοι και υποέλεγχο οι κίνδυνοι, αλλά οι θετικές αυτές πτυχές δεν πρέπει να μας κάνουν να την ανάγκη για πιο σταθερή και πιο καλά διαρθρωμένη οικονομική ανάπτυξη. Η υψηλή παραγωγικότητα λοιπόν ως παράγον της ανάπτυξης είναι απαραίτητη, χρειάζεται ως εκ τούτου καινοτομία. Οι διαθροτικές μεταρρυθμίσεις έχουν ουσιώδη ρόλο για τη δημιουργία του επιχειρηματικού εκείνου πλαισίου το οποίο, και περιβάλλοντος το οποίο θα οδηγήσει και στην καινοτομία. Και βέβαια σε αυτό έρχεται να ενωθεί και το κανονιστικό περιβάλλον σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορούν να συμβάλλουν οι σχετικές πρωτοβουλίες. Ε, πρέπει να έχουμε μια οικονομική και νοσηματική ένωση ε, αποδοτική και ευημερούσα και αυτό θα το καταφέρουμε με ένα καλό κανονιστικό πλαίσιο. Επομένως, πρέπει να ενισχύσουμε την καινοτομία. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να το πράξουμε αυτό που χρειάζεται και στην ε, λειτουργία τη Ευρωπαϊκής Νοσηματικής ένωσης Οικονομική και Ένωση και βεβαίως ε, προσβλέπω στη συζήτηση που θα ξεκινήσει από το έγγραφο σκέψεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενίσχυση της ΟΝΕ. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Είμαι στη διάθεσή σας για όποιε ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Thank you, President Draghi, uh, for your... Ευχαριστούμε κύριε Τράγκη για την πολύ πλούσια σε περιεχόμενο εισαγωγική ομιλία σας. Είναι μια ανάλυση βαθιά τη καινοτομία στον τομέα της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής τεχνολογίας, fintech, και νομίζω ότι αυτό το θέμα στην ουσία ευθυγραμμίζεται με τα ζητήματα που μας απασχόλουν. Ξεκινούμε με τον κύριο Brian Hayes ως πρώτο μιλητή τις ερωτήσεις. Ευχαριστώ Πρόεδρε Δράγκη, καλώς ήρθατε και πάλι στην ΕΚΟΝ. Είναι πολύ ενθαρρυντικό που ακούω τις παρατηρήσεις σας για το FinTech καθώς το θέμα αυτό πρόσφατα πέρασε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εσείς μας κάνατε παρατηρήσει σχετικά με τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που προβάλλονται. Έχω δύο ερωτήσεις. Η πρώτη έχει να κάνει ε, με το Brexit και συγκεκριμένο με τις τράπεζες οι οποίες ε, επανεγκαθίσταται από το Ηνωμένο Βασίλειο μεταφέρονται στην ε, Ευρωζώνη. Ε, η ECB είναι, είναι η τελευταία που θα αποφασίσει για το αν θα διοθωτήσει αυτές τις τράπεζες ε, να έρθουν εδώ. Έχετε σημαντικό ρόλο λοιπόν. Ο Ντάνιελ Νόιερ, ο συνάδελφός σας ε, και η ΕΣΜΑ και η ΟΠΑ μίλησαν ε, για τους, ε, τις εποπτικές αρχές στην Ευρωζώνη που δεν δημιουργούν, ένα, ε, δεν δημιουργούν ίσους όρους. Τι θα κάνει λοιπόν η ΕΚΤ σε αυτό το θέμα σχετικά με το πώς ε, ε, θα ρυθμιστεί η κατάσταση στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία θα πάνε αυτές οι τράπεζες. Τι θα κάνει εκεί η ΕΚΤ. Και η δεύτερη ερώτηση είναι Ιρλανδικής ε, φύσεως. Αν, από ό,τι ξέρετε, είχαμε μία κρίση στο τραπεζικό μας τομέα και μία από τις τράπεζες μας, η Αλενταέρ, είναι μία από τις 25 συστημικά, συστημικές τράπεζες σύμφωνα με τις δραστηριότητες της ΕΚΤ είναι μία από αυτές που είχε ε, πρόβλημα και η κυβέρνησή μας θέλει εν μέρη να την πουλήσει. Θεωρείτε λοιπόν ότι τώρα ήρθε η ώρα για να πουληθεί εν μέρη η τράπεζα αυτή και από τη δική σας πλευρά ποια θα ήταν τα μακροπρόθεσμα ωφέλη ενός καλύτερου και πιο σταθερού περιβάλλοντος τραπεζικού για τους Ιρλανδούς αλλά και γενικά για τη σταθερότητα του Ιρλανδικού τραπεζικού συστήματος. Ευχαριστώ για την πρώτη σας ερώτηση, ο κύριος Δράγκη. Φυσικά, η έκτε εσωτερικά προετοιμάζεται για κάθε περιπλοκή που μπορεί να προκύψει από το Brexit και αυτό φυσικά έχει να κάνει και με την εποπτική διάσταση. Οι τράπεζες ετοιμάζονται λοιπόν για την αποχώρηση της, του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση σταδιακά. Είμαστε σε επαφή και παρακολουθούμε εκ του σε αυτή τη διαδικασία. Όμως, όπως είπατε, αυτό δεν εξαρτάται μόνο από εμά, αλλά και από τις εθνικές αρμόδιες αρχές. Φυσικά, Είμαστε έτοιμοι να υποστηρίξουμε τις τράπεζες ώστε να, να αναδιοργανώσουν τις δραστηριότητες τους ε, στην περιοχή της ε, Ευρωζώνης. Είναι πολύ σημαντικό οι τράπεζες αυτές να έχουν προετοιμαστεί εγκαίρως. Το να είναι έγκαιρη η προετοιμασία είναι πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, ε, αυτό το έχω πει πολλές φορές, αλλά το ξαναλέω, πολλοί από τους κινδύνους ε, του Brexit έχουν να κάνουν με τον τρόπο που θα διαχειριστούμε αυτή τη διαδικασία. Εν ε, αν χειριστούμε σωστά την κατάσταση, πολλοί από αυτούς τους κινδύνους δεν θα υλοποιηθούν. Ε, είναι κάποια πράγματα τα οποία οι ίδιες οι τράπεζες πρέπει να κάνουν, να προετοιμαστούν εγκαίρως. Πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε ότι όλες οι τράπεζες που λειτουργούν στην ε, Ευρωζώνη ε, τηρούν τα πρότυπα της εποπτείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό έχει να κάνει όχι μόνο με την ασφάλεια και την σταθερότητα του συστήματος, έχει να κάνει με το κατά πόσο θα υπάρξει επιδείνωση ή όχι μετά τη διαδικασία αποχώρησης. Ε, υπάρχει ο κίνδυνος ενός κενού ή κατακαιρματισμού της εποπτείας. Ε, ε, κάτι που ως τώρα δεν μπορούμε ε, να αντιμετωπίσουμε με τον SSM. Υπάρχουν υποκαταστήματα σε τρίτες χώρες που δεν μπορούν να υποπληθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο εσείς λοιπόν ως νομοθέτες θα πρέπει να δράσετε σε αυτό το επίπεδο ώστε να διασφαλίσετε ότι οι ίδιοι κίνδυνοι αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο και ότι αποφεύγεται το ρυθμιστικό αρμπιτράζ που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα για το δεύτερο ερώτημά σας να πω ότι εξαρτάται αποκλειστικά από την Ιρλανδική κυβέρνηση ε, Γενικά να πω ότι καλό είναι τα οι κίνδυνοι να πάνε από τους φορολογούμενους στον ε, ιδιωτικό τομέα όταν μιλάμε για τις μετοχές τραπεζών. Η κατάσταση στις Ιρλανδικές ε, τράπεζες έχει προχωρήσει σημαντικά. Υπάρχει μεγάλη πρόοδος από την περίοδο της κρίσης και μετά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ που θέσατε και το θέμα της κούρσας προς τα κάτω και των broker deals είμαστε σε επαφή με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ε, και με τις εθνικές αρχές για να αντιμετωπίσουμε αυτό τον κίνδυνο η Περβόνς Πέρες έχει το λόγο ναι, δεν ξέρω αν είναι ένα καλό παράδειγμα αλλά θα θέσω κι εγώ δύο ερωτήματα όπως ο προηγούμενος ε, ομιλητής ε, κύριε Πρόεδρε έχετε συντάξει μαζί με άλλους τέσσερα άτομα την ε, έκθεση των πέντε προέδρων που είναι ξανά στην επικαιρότητα όπως βλέπετε. Επίσης είχατε πει ότι σε ό,τι αφορά τη λειτουργία της Οικονομικής και Ένωσης το θεσμικό ζήτημα θα πρέπει κάποια στιγμή να τεθεί. Διαπιστώνουμε όμως ότι εμφανίζονται κάποιες ιδέες αλλά κατακαιρματισμένες. Ε, ο, ο μηχανισμός ε, σταθερότητας να, ανατραπεί σε ένα ταμείο εκτός κοινοτικής λογικής και σε μια λογική πιο διακυβερνητική. Το πνεύμα της έξι των πέντε προέδρων όμως ε, ε, συνάδει με αυτή την προσέγγιση. Αυτή η προσέγγιση θα βοηθήσει την Οικονομική Νομισματική Ένωση να λειτουργήσει καλύτερα. Ε, αφενός έχουμε μια νομισματική πολιτική ε, εξαιρετικά ε, ολοκληρωμένη, ενώ στη δημοσιονομικό επίπεδο τα κράτη-μέλη είναι αυτά τα οποία έχουν τον πρώτο λόγο. Το δεύτερο ερώτημά μου τώρα έχει να κάνει με το την νομισματική πολιτική της Ένωσης και το μέλλον της. Έχετε αναλάβει κάποιες δεσμεύσεις στο τέλος του έτους. Ε, τώρα υπάρχουν διαφορετικές ε, εκτιμήσεις σε ό,τι αφορά ε, την επικοινωνιακή πολιτική σας για το τι θα συμβεί μετά το τέλος του έτους. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την εξέλιξη των μισθών. Στο Βερολίνο την περασμένη εβδομάδα Ακούσαμε ότι ήδη από τον Ιούνιο υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ε, για τους μισθούς ε, που μας δίνουν μια εικόνα για το πώς θα βγούμε από αυτή την νομισματική πολιτική που ακολουθείται αυτή τη στιγμή. Μπορείτε να μας πείτε κάτι περισσότερο σήμερα επ' αυτού. Ναι, ευχαριστώ. Ακούστε, συμφωνώ μαζί σας, ε, δεν θα έπρεπε βέβαια να το πω, διότι έχω ε, συντάξει αυτό το κείμενο μαζί με άλλους τέσσερις. Ε, είναι μια πρώτη απόπειρα για να σχεδιάσουμε τι θα συμβεί στο μέλλον. Οπότε εξετάζουμε δύο διαφορετικούς ορίζοντες. Τι θα γίνει βραχυπρόθεσμα και τι θα γίνει μακροπρόθεσμα. Η αλλαγή σε ό,τι αφορά τον σκοπό του ESM είναι πιο μακροπρόθεσμο ζήτημα. Διότι θα πρέπει να αλλάξει η συνθήκη. Εν πάση περιπτώσει, είναι πάρα πολύ νωρί να σας, για να σας πω εγώ κάτι συγκεκριμένο επ' αυτού. Θα πρέπει να το μελετήσουμε περαιτέρω. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι να μην έχουμε μια προσέγγιση κατακρεματισμένη. Να μπορέσουμε συλλογικά να καθορίσουμε, να ορίσουμε ποιον δρόμο θέλουμε να ακολουθήσουμε. Έναν δρόμο που θα μας οδηγήσει προς μία σύγκληση. Μία σύγκληση που θα βασίζεται στην ε, δημιουργία δυνατοτήτων σε θεσμικό επίπεδο και όχι σε κανόνες μόνο. Πρέπει να έχουμε λοιπόν ένα κοινό δρόμο που θα ακολουθούμε όλοι μαζί και όχι μια προσέγγιση à la carte. Τώρα, για την νομισματική πολιτική. Όπως ξέρετε θα έχουμε ε, μια συνάντηση του Συμβουλίου την ερχόμενη εβδομάδα, τον, τον των ε, Κυβερνητών. Ε, αυτό που έχουμε δει ως τώρα, και όπως είπα και στην εισαγωγή μου, είναι ότι ενώ έχουμε βελτίωση της κατάστασης ό,τι αφορά την ανάπτυξη, ενώ όντως η ανάκαμψη είναι σταθερή, βασίζεται όλο και περισσότερο στην κατανάλωση και όχι τόσο στις εξαγωγές και είναι αρκετά διευρυμένη, αφορά πλέον πολλές χώρες και πολλούς τομείς. Εμείς, ε, σε ό,τι αφορά την διεύρυνση της ανάκαμψης, ε, έχουμε έναν δείκτη στον οποίο αναφερόμαστε που έχει να κάνει με την ανάπτυξη και την προσθέμενη αξία αυτής της ανάπτυξης στις διάφορες χώρες. Όσο λιγότερο κατακαιρματισμένος είναι αυτός ο δείκτης, τόσο ευρύτερη είναι και η διεύρυνση. Όσο... Ε, και βλέπουμε ότι ο δείκτης αυτό σήμερα είναι στο ίδιο επίπεδο με το 1997 δηλαδή πολύ πριν από την κρίση. Αυτό μας λέει κατά κάποιο τρόπο ότι πολλά τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε με την κρίση, ο χρηματοοικονομικός κατακαιρματισμός, η ανισομερής ανάπτυξη ε, σε διάφορες χώρες της Ευρωζώνης ε, είναι προβλήματα τα οποία αφήνουμε πίσω μας. Ταυτόχρονα, όταν βλέπουμε τι γίνεται σε επίπεδο πληθωρισμού, διαπιστώνουμε ότι ο πληθωρισμός που υποβόσκει είναι σε, χαμηλές, σε χαμηλό επίπεδο. Όμως ε, δεν σημαίνει το ίδιο με τον πληθωρισμό των εμφανή. Ένας από τους λόγους πάντως της, ε, του ελέγχου της, του πληθωρισμού είναι ότι είναι περιορισμένη και η αύξηση των μισθών. Βεβαίω, σιγά σιγά διαπιστώνουμε μια αύξηση ε, και στις τιμές παραγωγού και στους μισθούς σε κάποιους τομείς και σε κάποιες χώρες, αλλά είναι πολύ νωρίς για να μπορούμε ήδη να μιλήσουμε για αλλαγή στην ορισματική πολιτική μας. Δηλαδή οι προβολές που έχουμε αυτή τη στιγμή ε, μας οδηγούν στο να παραμείνει σαν νομισματική πολιτική εξαιρετική στήριξη Ο Νότης Μαριάς έχει το λόγο, παρακαλώ. Κύριε Ντράγκη, κύριε Ντράγκη, πότε και υπό ποιε προϋποθέσεις θα αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την ένταξη της Ελλάδας στην ποσοτική χαλάρωση, στο QE, προκειμένου να αρχίσει εκ μέρους του ευρωσυστήματος η αγορά ομολόγων του ελληνικού δημοσίου στο πλαίσιο του προγράμματος PSPP. Δεύτερον, η Τράπεζα της Ελλάδος στα έτη 2015 και 2016 έχει δαπανίσει στο πλαίσιο του QE 42,5 δισεκατομμύρια ευρώ για αγορά ομολόγων διεθνών υπερεθνικών οργανισμών. Υπό ποιε προϋποθέσεις θα μπορούσε να αγοράσει η Τράπεζα της Ελλάδος στο πλαίσιο του προγράμματος CBPP3 εταιρικά ομόλογα ελληνικών επιχειρήσεων και ομόλογα ελληνικών τραπεζών στηρίζοντας έτσι την ανάπτυξη στην Ελλάδα και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Επιπλέον, κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας θέσω υπόψη την παρακάτω πρόταση αναφορικά με τον τρόπο άσκησης νομισματικής πολιτικής στην Ευρωζώνη, πρόταση που κατέθεσα στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο στις 17 Μαΐου. Θα μπορούσε άραγε, κύριε Ντράγκη, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών να γίνει πιο ευέλικτο και πιο αποκεντρωμένο, ώστε η Εθνική Κεντρική Τράπεζα κάθε κράτους μέλους της Ευρωζώνης να μπορεί να ασκεί νομισματική πολιτική προσαρμοσμένη στις ανάγκες της οικονομίας του δικού της κράτους, αξιοποιώντας σε εργαλεία σειρά μη συμβατικών μέτρων νομισματικής πολιτικής, όπως είναι η ποσοτική χαλάρωση, μέχρι του ποσοστού συμμετοχής της εν λόγω κεντρικής τράπεζας στο κεφάλαιο της ΕΚΤ και ανάλογα με το ύψος του τρέχοντος ισολογισμού του ευρωσυστήματος. Δηλαδή πρακτικά για την Ελλάδα θα μπορούσε η Τράπεζα της Ελλάδος αξιοποιώντας το QE να ασκεί νομισματική πολιτική προσαρμοσμένη στις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας, δημιουργώντας χρήμα, creating money, μέχρι 70 δισεκατομμύρια ευρώ, όσο δηλαδή είναι το ποσοστό 2% που κατέχει η Τράπεζα της Ελλάδος στο κεφάλαιο της ΕΚΤ, εν ώψη του ότι ο ισολογισμός του ευρωσυστήματος είναι 3,5 εκατομμύρια ευρώ αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ. Thank you. Σας ευχαριστώ. Η απάντηση στην πρώτη σας ερώτηση είναι εξής. Αυτό που χρειάζεται είναι καταρχάς θετική κατάληξη της τρέχουσας διαπραγμάτευσης και βεβαίως χαίρομαι ιδιαίτερως για την συμφωνία που επετέφθη σε τεχνικό επίπεδο και λυπούμαστε που δεν υπάρχει σαφής ορισμός μέτρων για το δάνειο από το τελευταίο Eurogroup, για το χρέος. Βέβαια θα γίνει μετά η αξιολόγηση της βιωσιμότητας του χρέους από τους λοιπούς φορείς και θεσμούς, όμως χρειάζεται μια βιωσιμότητα χρέους που να επιτρέπει στην ΕΚΤ και το Διοικητικό Συμβούλιο σε απόλυτη ανεξαρτησία να ε, αξιολογήσουν. Και αυτό σημαίνει ότι και με αντίξωα σενάρια θα παραμένει βιώσιμο το χρέο. Και πάνω σε αυτό θα γίνει η αξιολόγησή μας με βάση τα σενάρια, αξιολόγηση κινδύνου, όπως είπαμε επανειλημμένως. Ας γίνει πρώτα συμφωνία λοιπόν, ας υπάρξει μια πλήρη συμφωνία και να βρεθούν μέτρα, τα μέτρα εκείνα τα οποία θα καταστήσουν βιώσιμο το χρέος, μακροπρόθεσμα. Η δεύτερη σας πρόταση. Αν ήταν να έχουμε 19 κεντρικέ τράπεζε με 19 διαφορετικέ νομισματικέ πολιτικέ, θα είχαμε και 19 διαφορετικά εθνικά νομίσματα. Ακριβώ εκεί έρχεται το ένα νόμισμα, στη μία νομισματική πολιτική. Όλοι μα οι στόχοι προσδιορίζονται ω στόχοι για ολόκληρη την Ευρωζώνη, όχι στόχοι για ένα συγκεκριμένο κράτο. Όταν, παραδείγματι, μιλούμε για πληθωρισμό, αναφερόμαστε σε πληθωρισμό για όλη την Ευρωζώνη και όχι για πληθωρισμό για μία χώρα έναντι μια αλλη Ευχαριστώ. Η πρότασή μου ήταν συγκεκριμένη. Σας ρώτησα για την Τράπεζα της Ελλάδος. Η Τράπεζα της Ελλάδος στο πλαίσιο του QE δαπάνησε 42,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Το ερώτημα είναι υπό ποιου όρους η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί να αγοράσει εταιρικά ομόλογα ελληνικών επιχειρήσεων και ομόλογα ελληνικών τραπεζών στο πλαίσιο του QE. If and when. Εάν και όταν επεκταθεί το QE, η ποσοτική χαλάρωση και στην Ελλάδα, θα έχουμε επιλεξιμότητα οποιασδήποτε ελληνικής επιχείρησης μέσα στο πρόγραμμα αγοράς εταιρικών ομολόγων εφόσον αυτές πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας όπως αυτά έχουν οριστεί για το πρόγραμμα. Ραμόν Τρεμόζα. Ραμόν Τρεμόζα. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ευχαριστώ κύριε Ντράκη. Καλώ ήρθατε για μια φορά. Έχω μια ερώτηση σχέση με τη διαφάνεια. Από το 2016 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει αγοράσει πάνω από 75 δισεκατομμύρια ευρώ αξία ομολόγων από δυτικέ επιχειρήσει με το σύστημα αγορά αγοράς ε, εταιρικών ομολόγων. Εγώ από την αρχή είχα τι επιφυλάξει μου, μου γιατί διαχέουμε έτσι τον κίνδυνο σε ευρωπαϊκέ επιχειρήσει και βεβαίω η αδιαφάνεια καθιστά ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Στη Γερμανία έχουμε βέλτιστε πρακτικέ τη Bundesbank, η οποία δημοσιεύει τα ονόματα των εταιριών αυτών τουλάχιστον. Αλλά δεν συμβαίνει το ίδιο με ορισμένε ε, κεντρικές τράπεζες των νότιων χωρών της ε, Ευρωζώνης, άρα δεν είναι δυνατόν να μάθουμε ούτε πιανών εταιριών τα ομόλογα, αλλά ούτε ποιος όγκος ομολόγων αγοράζεται. Έτσι λοιπόν, μαζί με πολλούς ευρωβουλευτές της Επιτροπής μας ζητήσαμε από την ΕΚΤ διευκρινήσεις σε σχέση με το πρόγραμμα αυτό, με μια σειρά ερωτήσεων που σας έχουμε αποστείλει, πριν από δύο εβδομάδες συγκεκριμένα. Θεωρούμε λοιπόν ότι αυτή η απουσία διαφάνειας σε επίπεδο κεντρικής τράπεζας παραβλάπτει την ΕΚΤ και είναι κρίμα αυτό, διότι η ΕΚΤ έχει κάνει μεγάλα βήματα προς τη διαφάνεια, όπως τη δημοσιοποίηση των γνωμών, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλα ζητήματα, τα οποία και εγώ έχω υποστηρίξει εδώ και πολλά χρόνια στο Κοινοβούλιο, που δείχνουν ότι όσο πιο μεγάλη είναι η διαφάνεια, τόσο πιο ισχυρή είναι η ΕΚΤ σε σχέση με το ευρύτερο κοινό. Γι' αυτό λοιπόν ερωτώ εάν η ΕΚΤ πρόκειται να υιοθετήσει και να δημοσιεύσει κατευθυντήριες γραμμές για περισσότερη διαφάνεια στο πρόγραμμα ESPP. Ευχαριστώ. Θα πάρετε και γραπτή απάντηση στην ερώτησή σας, γιατί ήταν γραπτή και η ερώτησή σας. Αλλά παρόλα αυτά να πω κάποια πράγματα στο στάδιο αυτό. Έχουμε έξι εθνικές κεντρικές τράπεζες οι οποίες ε, λαμβάνουν μέρος σε αυτό το πρόγραμμα και όντως δημοσιεύουν μία ε, λίστα με τις μετοχές που έχουν σε ESPP ε, που μπορεί να ε, χρησιμοποιηθούν για δανεισμό χρεογράφων. Μπορεί κανείς λοιπόν να βρει τις πληροφορίες μέσα από τα δεδομένα που δίνουν οι τράπεζες αυτές ε, μέσω της αγοράς αλλά και από το κεντρική πύλη της ΕΚΤ. Μπορεί να γίνει online αναζήτηση αυτών των πληροφοριών που θα δείξει και τον εκδότη ε, των ομολόγων. Κάθε εθνική κεντρική τράπεζα που αγοράζει τα ομόλογα αυτά ε, μπορεί, με τη, έχει τη διακριτική ευχέρεια να αναφέρει αυτά τα στοιχεία μαζί με τα ESIN στοιχεία. Οι πληροφορίες που παρέχει η ΕΚΤ είναι αρκετές. Δεν νομίζουμε ότι υπάρχει λόγος να γίνει πιο κεντρική η δημοσίευση που αυτή τη στιγμή είναι στα χέρια πλήρως, στα χέρια των εθνικών κρατών κεντρικών τραπεζών, αλλά θα πάρετε και περαιτέρω γραπτές πληροφορίες με την γραπτή ε, απάντηση που θα σας δώσουμε. Μια επερώτηση. Κύριε Πρόεδρε Τράγκη, χωρίς επαρκή διαφάνεια υπάρχει ο κίνδυνος ε, κακής χρήσης ε, της νομισματικής πολιτικής από κάποιες κεντρικές τράπεζες για να μπορέσουν να αποφασίσουν για τον καπιταλισμό. Ας πούμε στην Ισπανία μόνο τρεις είναι οι εταιρείε οι οποίες πήραν πάνω από το 50% όλων των εξαγορών που έγιναν στην Ισπανία σύμφωνα με τα δημοσιεύματα. Νομίζω λοιπόν ότι αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να είναι συγκεντρωμένα σε επίπεδο έκτα και να προέρχονται από όλες τις ευρωπαϊκές, από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες, διότι αλλιώς είναι business as usual. Προσπαθούμε εμείς να δικαιολογήσουμε στο εκλογή, στους εκλογείς μας ε, πράγματα που έχουν να κάνουν με την πειθαρχία της αγοράς. Ε, δηλαδή, εμείς τροφοδοτούμε ε, εταιρείες οι οποίες είναι βιώσιμες στην αγορά ή όχι. Απάντηση. Να σας διαβεβαιώσω ότι οι εταιρείε επιλέγονται με βάση κριτήρια επιλεξιμότητας κινδύνου. Ε, δεν υπάρχει κάποια πρόθεση να ευνοήσουμε τη μία εταιρεία ή την άλλη. Υπάρχουν κάποιες κατευθυντήριες γραμμές ε, και κάποια στοιχεία που μαζί με την ΕΚΤ αποφασίζουν οι Εθνικές Κεντρικές ε, Τράπεζες. Δεν θα σας αποκαλύψουμε ούτε τον όγκο, ούτε τις κατευθυντήριες γραμμές, διότι ε, αν αυτό γίνει θα υπάρχουν οι άνθρωποι στην αγορά που θα ε, εμποδίσουν το έργο μας. Ε, πότε θα τελειώσει αυτό. Δεν προβλέπεται. Είναι ένα συνεχές πρόγραμμα. Είναι σαν αυτό που είπα πριν. Είναι η στάση μας σε επίπεδο νομισματικής πολιτικής. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει. Ευχαριστούμε. Μικέλ Ούρμπαν Κρέσπο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Ντράγκη, το ζήτημα της, τραπεζ... της διάσωσης των τραπεζών εξακολουθεί να είναι στην πολιτική αλλά και δικαστική επικαιρότητα της χώρας μου. Όπως γνωρίζετε, ο εξωτερικός ελεγκτής Deloitte ε, του υπευλήθη ένα πρόστιμο για το ρόλο του στον έλεγχο της Μπάνκια πριν από την ε, διάσωση. Είχε κάνει 12 σαφή λάθη που έκρυβαν τι πραγματικές απώλειες της Μπάνκια. Στις τελευταίε εβδομάδες ο δικαστής μάλιστα απέκλει κατηγορίες σε έναν από τους συνεργάτες της Deloitte για την ε, εισαγωγή στο χρηματιστήριο της Μπάνκια και συνεχίζεται ε, η κατηγορία εκπέμπτη στην ίδια την εταιρεία για, σε επίπεδο αστική ευθύνη. Είναι γνωστό ότι ο Ροντρίγκο Ράτο όταν ήταν πρόεδρος τη Μπάνκια σύναψε συμβόλαια με, τον, με, την, με την Λέζαρντ που είναι άλλο εξωτερικό ελεγκτή, ενώ ταυτόχρονα λάμβανε χρήματα από αυτή την εταιρεία σε έναν λογαριασμό στο εξωτερικό. Δυστυχώ αυτό που συμβαίνει στη χώρα μου συμβαίνει και αλλού, σε όλη την Ευρώπη. Είναι ένα πραγματικό ε, πλιάτσικο που γίνεται από τι τέσσερι μεγάλε ε, εταιρείε ελέγχου ε, και βλέπουμε ότι οι μεταρρυθμίσεις της νομοθεσίας υποχρεώνουν μόνο αλλαγή του, λεκτικού, του εξωτερικού ελεκτή κάθε, κάθε, κάθε, 10 χρόνια. Τι μπορεί λοιπόν να κάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως ε, εποπτική υπεύθυνη αρχή για να σταματήσει αυτή η κατάσταση ολιγοπολίου και να μην οδηγούμαστε σε πρακτικές που διέπονται από διαφάνεια και απάτη. Έχετε σκεφτεί τη δημιουργία ενός εξωτερικού ελεκτή δημόσιου ανεξάρτητου έτσι ώστε να μην υπάρχει εξάρτηση από τον ιδιωτικό τομέα και από το παρόν ολιγοπόλιο. Ευχαριστώ. Thank you. Uh, now, won't comment on specific... Ναι, ένα σχόλιο. Ε, δεν σχολιάζω μάλλον για επιμέρους ε, εταιρείε και όργανα. Θα σας δώσω γραπτός μια απάντηση, διότι αυτή τη στιγμή, για μένα τουλάχιστον, για μένα δεν είναι σαφές ποιος επιλέγει τους εξωτερικούς ελεγκτές και ποια είναι η διαδικασία επιλογής. Τους διαλέγει ε, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η, το σκέλος της Εποπτείας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η DigiComp και οι δύο είναι κάτι το οποίο θα μπορούσα να σας εξηγήσω καλύτερα εφόσον απαντήσω γραπτός στο ερώτημά σας. Η πρόταση ενός συνεξάρτητου δημόσιου ελεγκτή είναι μια ιδέα η οποία χρήζει εξέτασης. Αυτή τη στιγμή βεβαίως δεν έχω ούτε από αυτού κάποια άποψη. Ευχαριστώ. Thank you. Philip Lamberts. Ο Φίλιπ Λαμπέρτς έχει το λόγο. Καλό απόγευμα κύριε Πρόεδρε. Δύο ερωτήματα. Θα είμαι σύντομος για την Ευρωζώνη καταρχήν. Η νέα κατάσταση στη Γαλλία ενδεχομένως να δώσει κάποιες δυνατότητες. Θέλω να σας ρωτήσω, ε, να, αυτή η ιδέα ενός προπολογισμού της Ευρωζώνης με δυνατότητα δανεισμού ε, θεωρείτε ότι είναι κάτι που πρέπει να συμβεί, που θα ήταν καλό να συμβεί ή κάτι που δεν πρέπει να συμβεί έτσι ώστε να αγγιθούμε τη βιωσιμότητα του κοινού νομίσματος. Το δεύτερο ερώτημα έχει να κάνει με την μεταρρύθμιση της ε, ε, αγοράς εργασίας. Είναι κάτι που ζητούμε εδώ και καιρό, ζητούμε ελαστικοποίηση της αγοράς εργασίας, ε, όπως μεταρρυθμίσεις που έλαβαν χώρα στη Γερμανία κατά κάποιο τρόπο, υπό μάλιστα μια κυβέρνηση κοκκινοπράσινη, έτσι, στα τέλη της δεκαετίας του 90. Βλέπουμε ότι όταν αυξάνεται η απασχόληση, αυτό συμβαίνει με τέτοιο τρόπο όπου έχουμε κυρίως μερική απασχόληση. Ε, δεν είναι θέσεις απασχόληση μακράς διαρκείας, δεν θέλω να πω ότι όλες είναι κακές θέσεις εργασίας, αλλά σίγουρα δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ποιοτικέ εγώ δεν θέλω να μιλήσω για το ποσοστό ανεργία, θέλω να μιλήσω για το ποσοστό απασχόληση. Είναι στο 75% στη Σουηδία και μόλις 68% στη Γερμανία, 63% στο Βέλγιο, 55% στην Ιταλία. Μιλάμε μιλάω για την πλήρη απασχόληση. Και όταν βλέπουμε τη δυναμική με βάση τη αγορά εργασία με βάση αυτήν την, αυτό το πρίσμα, δεν υπάρχει κανένα δημοσιονάπτυξη που μπορεί να μα φέρει κοντά στην πλήρη απασχόληση. Ίσως λοιπόν οι διαθροτικές αλλαγές που χρειαζόμαστε για την αγορά εργασίας και τη σχετική πολιτική και αυτό βεβαίω συνδέεται και με τις δίπλα ε, των φορολογικών και της κοινωνικής πολιτικής ίσως να μην είναι τελικά αυτή που εσείς ευαγγελίζεστε. Θα ήθελα να ακούσω μια απάντηση από αυτό. Ναι, για το πρώτο. Ακούστε, είναι μια στιγμή ε, σκέψης. Είναι μια στιγμή πρέπει να αναλογιστούμε τι θα κάνουμε στο μέλλον. Να είναι σαφέστερα τα πράγματα και να βλέπουμε και πιο μακριά από το παρελθόν. Θα πρέπει λοιπόν τώρα να σκεφτούμε κατά πόσο οι κανόνες, το πλαίσιο σύγκλησης που έχουμε θεσπίσει Ε, κατά πόσο χρήζει βελτίωσης ή όχι. Η εμπειρία των τελευταίων ετών μας λέει ότι η Οικονομική γνωσματικη Ένωση άντεξε στην κρίση, αλλά βρέθηκε πολύ, πολύ κοντά σε πολύ κρίσιμες καταστάσεις. Είναι λοιπόν λογικό να ξανασκεφτούμε αυτό το οικοδόμημα έτσι ώστε να μην μπορεί να απειλείται τόσο συχνά και τόσο άμεσα όπως το παρελθόν. Έτσι λοιπόν η ΩΝΕ παραμένει εύθραυστη και πρέπει να ολοκληρωθεί. Γνωρίζουμε ότι μέρος του έθραυστου χαρακτήρα της είναι ότι δεν έχει ολοκληρωθεί και πρέπει λοιπόν να προχωρήσουμε. Πρέπει να προχωρήσουμε σε διάφορα επίπεδα είναι πολλά αυτά που μπορούμε να κάνουμε, μπορούμε να κάνουμε σύντομα, σε μικρό χρονικό διάστημα, κάποια άλλα θα πρέπει να τα σκεφτούμε πιο καλά. Δεν θα πρέπει να φοβόμαστε να αλλάξουμε τη συνθήκη, παραδείγματο χάρη, εφόσον χρειαστεί. να αρχίσουμε δηλαδή να σκεφτόμαστε το μέλλον χωρίς να δεσμευόμαστε από την υπάρχουσα συνθήκη. Και αυτό ήδη είναι πρώτο σημαντικό βήμα. Έχουμε πει πολλές φορές ότι να υπάρχει ε, μια δυνατότητα δημοσιονομική ε, είναι ένα σημαντικό, ένα σημαντικός παράγοντας για την ολοκλήρωση, ολοκλήρωση της Ένωσης. Έτσι θα μπορούσαμε να είμαστε πολύ πιο ανθεκτικοί απέναντι σε πιέσεις και σε κρίσεις σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης. Αν δούμε άλλωστε τι συμβαίνει ε, παντού, σε οποιαδήποτε τέτοιου είδους ένωση υπάρχει ένας προπολογισμό ομοσπονδιακό. Το θέμα είναι πώ θα φτάσουμε εκεί. Ένα προπολογισμό τη ίδια τη Ένωση. Το θέμα είναι λοιπόν πώ θα φτάσουμε εκεί και η απάντηση είναι αυτή που έχουμε πει και στο παρελθόν. Χρειάζεται πρώτα εμπιστοσύνη μεταξύ των χωρών, με εμπιστοσύνη και σύγκληση σύγκληση ε, διότι μια ετερογενής ένωση θα, είναι, θα ήταν εύθραυστη ε, από δομικής πλευράς. Για να υπάρξει λοιπόν σύγκληση θα πρέπει πρώτα να ολοκληρώσουμε αυτό που έχουμε σχεδιάσει έως τώρα αλλά χρειάζεται και σύγκληση σε επίπεδο πολιτικών σε επίπεδο μεγάλων σοβαρών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, ολοκλήρωσης τραπεζικής ένωσης, όλα αυτά αποτελούν μέρος της διαδικασίας σύγκλησης. Για να έρθω τώρα στο δεύτερο ερώτημά σας. Η μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας. Εγώ πιστεύω ότι λίγο πολύ, εντάξει βεβαίως είναι αλήθεια αυτό που είπατε, συχνά η αύξηση της απασχόλησης παρότι είναι σημαντική, μην ξεχνάμε έτσι, 5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν τα τέσσερα τελευταία χρόνια. Πολλές περισσότερες από ό,τι πριν από την κρίση. Και αυτό είναι θετικό. Βεβαίως, από την άλλη είναι αλήθεια ότι κάποιες από αυτές τις νέες θέσεις απασχόλησης δεν είναι καλής ποιότητας. Και αυτό είναι αλήθεια. Τώρα, τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Να σας πω επίσης ότι σε γενικές γραμμές τα περισσότερα κράτη-μέλη της Ένωσης έχουν προχωρήσει σε μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας τους για να τις καταστήσουν πιο ευέλικτες. Υπάρχει όμως τώρα ε, μια άλλη σειρά μεταρρυθμίσεων που πρέπει να λάβουν χώρα. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε μια κατάσταση όπου οι νέοι στην αγορά εργασίας θα έχουν τις απαραίτητες δεξιότητες έτσι ώστε να παραμείνουν στην αγορά εργασίας. Και για να αποκτήσουν αυτές τις δεξιότητες, εκεί είναι που χρειαζόμαστε μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Είναι και αυτό το σκέλος. Δηλαδή στο παρελθόν μπορούμε να έχουμε δώσει έμφαση στην ευελιξία. Σήμερα όμως πρέπει να δούμε πώς θα βελτιωθούν τα εκπαιδευτικά μας συστήματα έτσι ώστε να δημιουργούμε θέσεις εργασίας που να είναι ε, βιώσιμες, μακροπρόθεσμες αλλά και ποιοτικέ. Και αυτό πρέπει να συνοδεύεται βέβαιως και από αύξηση των μισθών. Διότι πάει από κοινού, πάει χέρι-χέρι με μία αύξηση της αγωνιστικότητας. Είναι δηλαδή μία κατάσταση όπου όλοι κερδίζουν. Ευχαριστώ. Δεν χρειάζεται να σας θυμίσω ότι αυτό το κοινοβούλιο, αυτή η επιτροπή έχει εγκρίνει έκθεση η οποία προτείνει από κοινού να προχωρήσουμε σε μεγαλύτερη σύγκληση έτσι ώστε να αντιμετωπίζουμε μελλοντικούς κραδασμούς. Ε, κάτι που είναι μια φιλόδοξη αλλά και ε, ρεαλιστική πρόταση. Ο κύριος Χάνεμανς. Συνήθως δίνεται μία τυπική απάντηση σε αυτό, αλλά θα το προσπαθήσω για άλλη μια φορά και θα σας ρωτήσω πότε θα σταματήσει η ποσοτική χαλάρωση, που νομίζω γιατί νομίζω ότι επηρεάζει αρνητικά τις καταθέσεις και τα συνταξιδοτικά ταμεία σε όλη την Ευρωζώνη. Η ΕΚΤ δεν είναι πολιτικό όργανο. Λέτε ότι εσείς είστε εδώ για να διασφαλίσετε τη σταθερότητα των τιμών, όμως άλλοι λένε πως έχετε τον πολιτικό στόχο έτσι ώστε ε, ε, να... Ε, Όμως το γεγονός είναι ότι τα 500 δις ε, στον προϋπολογισμό σας το είναι πολύ σημαντικό ποσό. Ένα ποσό ε, που δεν πρέπει να ξεπεράσει το 33% του κρατικού χρέους ε, ενός μέλους της Ευρωζώνης. Όταν σας ρώτησαν στο Ολλανδικό Κοινοβούλιο πρόσφατα για το γεγονός ότι ε, αν υπήρχε μια αποχώρηση, εσείς θα παίζατε πολιτικό ρόλο, όμω είπατε ότι δεν υπάρχει τέτοια πιθανότητα. Να το θέσω αλλιώς το ερώτημα. Αν έπρεπε να σεβαστείτε το 33% θα μπορούσατε να πείτε ποια είναι η, χώρα που θα έπρεπε να μειώσει το κρατικό της χρέος ως αποτέλεσμα αυτού, μέσα στα πλαίσια του προγράμματος της ποσοτικής χαλάρωσης φυσικά. Ευχαριστώ πολύ. Να πω αμέσως ότι γνωρίζουμε πως υπάρχει μια συνεχής κατάσταση με πολύ χαμηλά επιτόκια οποία στην ουσία αποτελεί πρόκληση κυρίως για τα συνταξιδοτικά ταμεία και τις ασφαλιστικές εταιρείες, αλλά κυρίως ε, και για τους καταθέτες γενικότερα. Και υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούν να γίνουν για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση σε επίπεδο καταθετών ασφαλιστικών και συνταξιδοτικών ταμείων. Η δράση που πρέπει να αναλυφθεί στην ουσία έχει αναλυφθεί ήδη. Παρ' όλα αυτά, ο λόγος που γίνεται αυτό, όπως το είπα πολλές φορές, είναι επειδή η κατάσταση θα, απαιτούσε ως προαπαιτούμενο δηλαδή αυτά τα χαμηλά επιτόκια έτσι ώστε για να γίνει ένα restart που τώρα αποδίδει. Οι λόγοι λοιπόν που πολλές φορές αναφέρονται από πολλές πλευρές για το πρόγραμμά μας ε, είναι κάτι που κάθε φορά το λέω στην απάντησή μου. Ο νόμος μας δεσμεύει για τη σταθερότητα των τιμών και να έχουμε έναν πληθωρισμό κάτω από το 2% και γι' αυτό δημιουργήσαμε αυτά τα προγράμματα εξαγοράς ε, κεφαλαίων. Και γι' αυτό αγοράζουμε και ομόλαγα τακτικά με έναν ρυθμό που φτάνει τα 60 δις ε, ευρώ το μήνα αυτή τη στιγμή. Και παρόλο που γνωρίζουμε τις παρενέργειες που μπορεί να έχουν αυτά τα προγράμματα, γνωρίζουμε ταυτόχρονα ότι μας δεσμεύει και η συνθήκη να μην κάνουμε νομισματική χρηματοδότηση. Και γι' αυτό έχουμε αυτά τα όρια για την έκδοση στο πρόγραμμά μας. Τούτου λεχθέντος και εφόσον συνεχίσει να ομαλά το πρόγραμμα, εμείς, το Διοικητικό Συμβούλιο, ποτέ δεν σχεδίαζε να παραβιάσει τα όρια που είναι εκεί και θα παραμείνουν εκεί. Και δεν είμαι σε θέση να απαντήσω στην ερώτησή σας ποιες χώρες θα αγοράζουν λιγότερα ε, ομόλογα για να μπορέσουν να σεβαστούν αυτά τα όρια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πέτριξ Πανστόρ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κύριε Ντράγκε. Στην αρχή του έτους ε, απαντήστε την απάντηση του συναδέλφου Άννη Ζάνη ε, μιλήσατε ε, στις 18 Ιανουαρίου και είπατε ότι αν μια χώρα έπρεπε να φύγει από το σύστημα του ευρώ, θα έπρεπε ε, να μπορέσουν πρώτα να ρυθμιστούν οι υποχρεώσεις στην Κεντρική Τράπεζα. Είναι μια απάντηση στο υποθετικό σενάριο μιας αποχώρησης από την Ευρωζώνη η αποχώρηση φυσικά είναι το worst case σενάριο, το χειρότερο σενάριο. Μιλάμε λοιπόν για τέτοια σενάρια ενδεχομένω ε, με εκπλήσει η απάντηση που δώσατε στο Ολλανδικό Κοινοβούλιο. Σας ρώτησαν τι γίνεται αν θέλει ένα μέλος της Ευρωζώνης να διαρθρώσει το χρέος του, όχι να βγει από την Ευρωζώνη, απλώς να αναδιορθώσει. Η απάντησή σας ήταν δεν θέλουμε να ε, σκεφτόμαστε την πιθανότητα πραγμάτων που δεν έχουν καμία πιθανότητα να συμβούν και, με ρωτήσατε, και ρωτήσατε μετά ενοχλημένος γιατί το ρωτάτε αυτό. Αυτή την ερώτηση σας θέτω και πάλι. Με βάση την απάντηση που δώσατε στην αρχή, στις αρχές Ιανουαρίου στο συνάδελφο για ένα υποθετικό σενάριο, ε, το χειρότερο σενάριο. Σας ρωτάω λοιπόν τι θα γίνει αν ένα μέλος της Ευρωζώνης είναι αφαιρέγγιο και πρέπει να αναδιαρθρώσει το χρέος του ειδικότερα ε, όταν μιλάμε για μεγάλα ποσά που βρίσκονται στο προϋπολογισμό σε δάνεια. Και φυσικά η ΕΚΤ δεν θα κάνει το ίδιο όπως το 2010 όταν ήταν πρώτων θυρών της χρεοκοπίας η Ελλάδα που αγόρασε αυτά τα κρατικά ομόλογα έτσι ώστε να αλλάξει αυτή η πτώχευση, η πορεία προς την πτώχευση. Now, let να σας δώσω δύο-τρεις γρήγορες απαντήσεις. Καταρχάς, να πω ότι το ευρώ ε, δεν ανακαλείται. Τα θέματα αυτά ε, για, ε, για το παθητικό του στόχου 2 δεν τα επαναλαμβάνω. Τώρα, τι θα γίνει αν ένα κυρίαρχο κράτος αναδιαρθρώσει το χρέος του. Απάντηση, κοιτάξτε στην Ελλάδα. Την Ελλάδα. Τρίτον, Είπατε ότι φέρουμε τον κίνδυνο για όλη την Ευρωζώνη εξαιτία των ομογολόγων που αγόρασε η έκτε στι διάφορε χώρε. Δεν υπάρχει επιμερισμό κινδύνων, μόνο σε περιορισμένο ποσοστό. Σε μεγάλο βαθμό, λοιπόν, ο κίνδυνο αναδιάρθρωση χρέου ε, ε, είναι ένα κίνδυνο που φέρουν οι κεντρικέ τράπεζε, εθνικέ τράπεζε. Ευχαριστώ, ο Μάρκου Φέμπερ. Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ να αναφερθώ στην Τάγες Zeitung, ίσως να ήταν πολύ πιο ανώδυνο αυτό. Έχουμε ένα ρεκόρ λοιπόν το Μάρτιο. Τέσσερα κράτη μαζί έχουν πλεόνασμα 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ μαζί με τη Γερμανία. Τρίλιον το λέμε στα αγγλικά από ό,τι ξέρω, επομένως είναι το 3 εκατομμύριο και στην Νότια Ευρώπη έχουμε σημαντικά ελλείμματα αντίστοιχα. Ερωτώ λοιπόν από τις εξελίξεις αυτές. Βλέπετε ότι μπορεί να είναι βιώσιμες. Την τελευταία φορά μας είχατε πει ότι έχουν σχέση με την προσωπική χαλάρωση τα φαινόμενα αυτά, αλλά και η Γαλλία θα έπρεπε να πούμε ότι έχει θετικό υπόλοιπο. Αυτό δεν το καταλαβαίνουμε λοιπόν πώς γίνεται και ρωτούμε εάν θεωρείτε ότι θα πρέπει να γυρίσουμε σε ένα σύστημα ίσως και όπως συνέβαινε πριν από την κρίση. Απάντηση. Ναι, ευχαριστώ. Καταρχάς θέλω να πω ότι ο στόχος, γιατί είναι τόσο διαφορετικό σε σχέση με αυτό που εμφανιζόταν το 2012, το 2013, στο χειρότερο σημείο της κρίσης δηλαδή. Εδώ έχουμε να κάνουμε με μια αποκεντρωμένη διαχείριση στην υλοποίηση της νομισματικής μας πολιτικής. Μεγάλο κομμάτι αυτού λοιπόν, αυτής της ανισότητας έχει να κάνει με το σύστημα αγοράς τίτλων. Και γιατί. Ας σημειώσουμε πρώτα το 80% των αντισυμβαλωμένων στις κεντρικές τράπεζες που πολλούν τα ομόλογα βρίσκονται έξω από τα σύνορα της χώρας την οποία έχει την έδρα της Κεντρική Τράπεζα. 50% των αντισυμβαλωμένων είναι εκτός της Ευρωζώνης, μάλιστα. Επομένως, ε, όταν η Κεντρική Τράπεζα μιας συγκεκριμένη χώρας αγοράζει ομόλογα από αντισυμβαλωμένους και αυτοί οι αντισυμβαλόμενοι μετά το ρευστό που παίρνουν το καταθέτουν όχι στην ίδια κεντρική τράπεζα που τους ε, αγόρασε τα ομόλογα, αλλά το χρησιμοποιούν ε, σαν κατάθεση σε κεντρική τράπεζα μεγάλων ε, χρηματοπιστωτικών κέντρων, κατά κύριο λόγο την Bundestag, Bundesbank. Εδώ λοιπόν έχουμε να κάνουμε με ένα target liability για την τράπεζα η οποία έχει πωλήσει τα ομόλογα και ένα target to asset για την Bundesbank ή την αντίστοιχη κεντρική τράπεζα που είναι στα μεγάλα χρηματοπιστωτικά κέντρα. Επομένως, το πρώτο ζήτημα είναι ότι έχουμε να κάνουμε με έναν αποκεντρωμένο τρόπο υλοποίησης της ε, πολιτικής εποπτείας. Δεύτερον, η πολιτική, αυτή η νομισματική πολιτική, πρέπει να δούμε πώς λειτουργεί στο σύστημα στην ε, εξασφάλιση αυτό που λέμε portfolio rebalance, ε, πανισοσκέλης του χαρτοφυλακίου. Δηλαδή, όταν αυτές οι τράπεζες χρησιμοποιούν τα έσοδα για να αγοράσουν άλλους τίτλους, ε, άλλο ενεργητικό ή άλλο τύπου ομόλογα, μέσα ή έξω από την Ευρωζώνη. Πρέπει λοιπόν όλες αυτές τις κινήσεις να τις παρακολουθούμε για να αντιληφθούμε ότι η αύξηση του target του liability σχετίζεται με την απώλεια ενδιαφέροντος από αυτούς που πολλούν τα συγκεκριμένα ομόλογα για τίτλους ενεργητικού της συγκεκριμένη χώρας. Και γιατί είναι διαφορετικό αυτό, η αύξηση δηλαδή στο target του liability που παρατηρήσαμε το 2012 και 2013. Οφειλόταν στο ότι οι τράπεζες στην Ευρωζώνη και ιδιαίτερα στην περιφέρεια στις περιφερειακές χώρες, είδαν ότι η χρηματοδότηση στηριζόμενη στην αγορά ε, εξαφανιζόταν και έπρεπε να στήσουν επαναχρηματοδότηση από την οικία κεντρική τράπεζα. Και αυτό ξεκίνησε, σε, οδήγησε σε σημαντική αύξηση του target του liability. Γιατί, διότι αυτές οι τράπεζες αναζητούσαν στοιχεία ενεργητικού από κεντρικές τράπεζες. Άρα έχουμε μια διαδικασία την οποία υποκινεί η ζήτηση σε εκείνη την περίοδο. Τώρα έχουμε μια διαδικασία την οποία ε, υποκινεί η προσφορά. Πολλούν δηλαδή ενεργητικό σε εμπορικές τράπεζες, στα εξωτικά ταμεία, ε, ταμιευτήρια, ασφαλιστές κτλ. Οι τράπεζες οι Και αποκεντρω... Γι' αυτό έχουμε ένα αποκεντρωμένο χαρακτήρα τη ε, νομισματική πολιτική σε σχέση με το higher target του liabilities. Υπάρχουν πιέσει, δείγματα πιέσεων στην αγορά. Όχι αυτή τη στιγμή. Εάν κοιτάξουμε του όρου τη χρηματοδότηση. είναι πολύ ευνοϊκή και για τις εμπορικές τραπέζε και για τι μη τραπεζικέ εταιρείε και για την πραγματική οικονομία εκεί όπου είναι πιεστικές οι συνθήκες το 2012 το 2013 μπορεί να είναι πάλι και βέβαια θα θυμάστε ότι ήταν πολύ ψηλά τα επιτόκια πολύ υψηλή δυσκολία εξασφάλισης χρηματοδότησης άρα η κατάσταση είναι κατ' ουσίαν πολύ διαφορετική από το 2012-2013 ως τώρα Ευχαριστώ Γιακόπ Φων Φάστσεκα. Πρόεδρε ευχαριστώ και χαίρομαι που σας βλέπω εδώ κύριε Ντράγκη δύο ερωτήσεις η πρώτη αφορά την προοπτική, όχι στο άμεσο μέλλον μεν, αλλά αργότερα, της αντιστροφής του, των τάσεων στο, στα επιτόκια. Μας δώσατε μια πολύ καλή εικόνα των προοπτικών, του ελέγχου των τιμών, αλλά θα ήταν καλό να κοιτάξουμε τι μπορεί να σημαίνει αντιστροφή των επιτοκίων και πάνω απ' όλα τι είδους πρόκληση μπορεί να φέρει για τις οικονομίες που έχουν χαμηλή ανάπτυξη. Και θέλω να ρωτήσω ποιες είναι οι πτυχές της συζήτησης που διεξάγεται τώρα ως προς την σοβαρή εμβάθυνση στην ε, Νομισματική Ένωση και πώς μπορούμε να προστατέψουμε από τέτοιου είδους κλειδονισμούς την ε, Νομισματική Ένωση. Πιο συγκεκριμένα, πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν προβλήματα που έχουν να κάνουν με τις κεντρικές τράπεζες. Και νομίζω ότι η απάντηση θα είναι ότι μπορεί να εξασφαλιστεί περισσότερη συνένεση για την ε, φορολογική ένωση με αυτό το επιχείρημα. Μια άλλη ερώτηση σε ένα θέμα που με ε, απασχολεί γιατί είναι η έκθεση που με τα CCP με το Brexit και τις σημαντικές προκλήσεις προς τον κανονισμό του χρηματοπιστωτικού τομέα που μπορεί σε ένα βαθμό να καλυφθεί με την ενίσχυση του καθεστώτος ε, ισοδυνάμου τρίτης χώρας, third country equivalence regime, ε, με την αναγνώριση της, ε, του Ηνωμένου Βασιλείου. Μετά έχουμε την εξοεδαφικότητα με την εποπτεία όπως την έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο εξωτερικό. Και το τρίτο θα ήταν ο επαναπατρισμός. Με ενδιαφέρει λοιπόν και αυτή είναι η ερώτησή μου ποιος από τους ε, τομείς ε, των ε, ελεγχόμενων κινδύνων για το χρηματοπιστωτικό κόσμο και κάθε χρηματοπιστωτικό τομέα χωριστά μπορεί να έχει μεγαλύτερη σημασία και θα πρέπει να σας απασχολήσει πιο άμεσα. Ευχαριστώ. Έχουμε ήδη δει αύξηση των επιτοκίων και η δική μας αξιολόγηση, η δική μας εκτίμηση είναι ότι αυτό οφείλεται ε, στην αύξηση των πραγματικών επιτοκίων αφενός και αφετέρου από την βελτίωση της οικονομικής κατάστασης ε, δηλαδή στην Ευρωζώνη. Αυτό είναι το πρώτο μέρος μάλλον και το δεύτερο μέρος έχει να κάνει με την ε, αύξηση της ασφα... του πριμ ασφάλισης δηλαδή για σε ό,τι αφορά την, τον αποπληθωρισμό δηλαδή υπάρχει αυτή η, η άποψη ότι ο αποπληθωρισμός δεν αποτελεί πλέον τόσο μεγάλο κίνδυνο, οπότε χρειάζεται μικρότερη ασφάλιση. Βεβαίω, στι τελευταίε 10-12 μήνε είχαμε μια μικρή αύξηση. Τώρα, αυτό έχει δημιουργήσει μια κατάσταση αστάθειας. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή. Μπορούμε να αποκλείσουμε ότι η αύξηση των επιτοκίων ε, θα οδηγήσει σε αστάθεια. Αυτό φυσικά και δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε. Είναι πάντως σαφές για να προσπαθήσω να απαντήσω την ερώτησή σας επί της ουσίας. Είναι σαφές ότι καθώς ο πληθωρισμός θα συγκλίνει προς το στόχο μας, καθώς αυτή η σύγκληση θα είναι πλέον ε, αυτόνομη, οι χώρες με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης θα, θα έχουν ε, υψηλό λογαριασμό σε επίπεδο επιτοκίων και θα πρέπει λοιπόν να έχουν τι κατάλληλε πολιτικέ για να το αντιμετωπίσουν αυτό και σε φορολογικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο ε, αύξησης, ενίσχυσης των ρυθμών ανάπτυξης. Αυτό είναι το πιο σημαντικό σκέλο της οικονομικής πολιτικής για αυτές τις χώρες. Τώρα, θα πρέπει να εξετάσουμε ε, κάποιο θεσμικό πλαίσιο που θα αποκλείει οποιαδήποτε αστάθεια ε, επειδή κάποιες χώρες έχουν μείνει πίσω στη διαδικασία σύγκλησης. Εάν δούμε βεβαίως την εμπειρία που έχουμε ιστορικά, στην αρχική φάση με τη συνθήκη του Μάστριχτ, αφενός οι χώρες πρέπει να δράσουν, να κάνουν αυτό που τους αναλογεί, να έχουν υγιείς δημοσιονομικές, οικονομικές πολιτικές, ταυτόχρονα, βεβαίως έχετε δίκιο, ε, πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα ασφάλισης, ένα, μια, ε, ένα απόθεμα και βεβαίως ε, σε θεσμικό επίπεδο πρέπει να ενδυναμώσουμε τους θεσμούς μας που, έτσι ώστε να είναι πιο ανθεκτικές απέναντι σε φαινόμενα αποσταθεροποίησης που προέρχονται από τις χώρες που έχουν μείνει πίσω. Και αυτό πρέπει να προχωρήσει. Είναι δηλαδή μια συνολική διαδικασία την οποία πρέπει να έχουμε κατά νου για το μέλλον. Τώρα για το δεύτερο ερώτημά σας. Θα ήθελα να αναφερθώ στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα CCPs που ε, δημοσιεύθηκε 4 Μαΐου και εκεί προβλέπεται μια σειρά από επιλογές για την βελτίωση του καθεστώτος εποπτείας ό,τι αφορά τα CCPs μεταξύ των οποίων και η ενισχυμένη εποπτεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και των απαιτήσεων. Αυτό βεβαίως ο Ευρωπαίος νομοθέτης θα τα αποφασίσει τελικά ποιο καθεστώς θα πρέπει να ακολουθηθεί ε, σε συστημικά σημαντικές εισηπείς των χωρών. Για μας, ε, ως Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, θα είναι σημαντικό, θα είναι κρίσιμο ε, να μπορέσουμε να διαφυλάξουμε το παρόν επίπεδο συμμετοχής σε ό,τι αφορά τη συστημική διαρκώς σημαντικές ε, δραστηριότητες που σχετίζονται με το ευρώ. Ανεξάρτητα από το πλαίσιο που θα αποφασίσει ο Ευρωπαίος νομοθέτης και από τη μορφή που θα πάρει η σχέση η Ευρωπαϊκή Ένωση του Βασιλείου στο μέλλον. Είναι πολύ νωρί, είναι πρόημο να γνωρίζουμε ποια θα είναι η τελική δομή. Αλλά αυτό που θέλουμε να διαφυλάξουμε τουλάχιστον είναι την παρούσα, το παρόν ε, επίπεδο συμμετοχής. Πρέπει να έχουμε λοιπόν τα κατάλληλα εργαλεία με βάση την ευρωπαϊκή νομοθεσία έτσι ώστε να μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι θα διαφυλάξουμε την σταθερότητα του νομίσματος ε, απέναντι στον ενδεχόμενο κίνδυνο ε, που δημιουργεί, ε, δημιουργούν οι offshore. Ε, και βεβαίως εδώ καλωσορίζουμε την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η ανακοίνωση αναγνωρίζει πλήρως τον ρόλο που πρέπει να παίζει η τράπεζα έκδοσης σε αυτό το νέο περιβάλλον. Ευχαριστώ, Γκαμπριέλ Μάτο έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, ευχαριστώ και τον κύριο Ντράγκη. Εγώ θα μιλήσω για το μέλλον. Το μέλλον της Ευρώπης ε, σε μια στιγμή αστάθειας και ε, αβεβαιότητας είπε η κυρία Μέκελ πριν από λίγο ότι έχει μείνει, έχει, είναι επίσημα σε η εποχή όπως να βασιστούμε σε άλλους πρέπει να βαστούμε στι δυνάμει μα. Αλλά και ο Γάλλο πρόεδρο είπε ότι το ευρώ δεν είναι πλήρε. Δεν μπορεί ε, να σταθεί χωρί σημαντικέ μεταρρυθμίσει. Έχω γίνει μια σειρά από προτάσει ε, που θα μπορούσαν να δεχτούν χώρε όπω η Ισπανία. Μια πιο ολοκληρωμένη φορολογική πολιτική, έναν υπουργό οικονομικών ε, Ευρωπαίων με εποπτεία κοινοβουλευτική και να προχωρήσει Τραπεζική Ένωση. Θα ήθελα, αν μπορείτε, να πείτε τη γνώμη σα για αυτέ τι προτάσει και αν θα μπορούσε να λειτουργήσει μια τέτοια ατζέντα. Επίσης, για το μέλλον των Ευρωπαϊκών Αρχών Εποπτείας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει μια δημόσια διαβούλευση για το μέλλον αυτών των οργανισμών για να δούμε κατά πόσο πληρούν τις προϋποθέσεις και κατά πόσο πετυχάνει το στόχο της διαφύλαξης του δημοσίου συμφέροντος. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε εσείς ποιο πιστεύετε πρέπει να είναι να είναι το μέλλον αυτών των φορέων. Και βεβαίω η κλασική ερώτηση που κάνω πάντα ε, και που βεβαίω την έχουμε όλοι, η αύξηση των επιτοκίων. Είπατε εσεί σαφώ κάτι το, με το συμφωνούμε όλοι, υπάρχει αύξηση τη ανάπτυξη, η ανεργία είναι πιο χαμηλή από το 2009, υπάρχει αύξηση τη εμπιστοσύνη τη αγορά. Ε, χρειάζονται βεβαίω ε, διαφορετικέ μεταρρυθμίσει με έμφαση στην καινοτομία, είπατε. Κάποιοι έχουν αλλάξει όμως την πολιτική τους, ε, η Federal Reserve, παραδείγματος χάρη, ό,τι αφορά τα επιτόκια. Εσείς ποια σενάρια έχετε κατά νου, ποια σενάρια έχει κατά νου η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και βεβαίως η ερώτηση του ενό εκατομμυρίου, ξέρω ότι θα απαντήσετε βέβαια, ε, υπάρχει περίπτωση αύξηση των επιτοκίων, να λάβει χώρα αύξηση των επιτοκίων εντό των επιμένων μηνών. Και τέλος, ε, η εμπορική μας σχέση με τις ΗΠΑ. Ο πρόεδρος Τραμπ ήταν αυτή την εβδομάδα εδώ στην Ευρώπη και ήταν, ήταν ισχυτικά αυτά που ακούσαμε, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την εμπορική πολιτική. Θα ήθελα να μου πείτε και από αυτού την άποψη, αν μπορείτε. Ευχαριστώ. Ε, thank you Ευχαριστώ. Καταρχάς να απαντήσω στην πρώτη σας ερώτηση. Σίγουρα καλωσορίζουμε τη διαδικασία διαβούλευσης που ξεκίνησε η, η Επιτροπή για το ρόλο των Ευρωπαϊκών ε, ε, Αρχών Σταθερότητας που είναι ακριβώς η αρχή για τη δημιουργία μιας ε, τραπεζικής ένωσης και ο πυλώνας στον οποίο θα δημιουργηθεί και η Ένωση Κεφαλαγοράς. Ε, είναι σίγουρο ότι καλό είναι να έχουμε ένα σύστημα ρύθμισης και εποπτείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη συγκεκριμένα. Έχουμε συνεργαστεί με την ε, Επιτροπή και με τις ε, Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές οι οποίες λειτουργούν εδώ και έξι χρόνια. Άρα ήρθε η ώρα να τις ε, ξανακοιτάξουμε, να τις αναθεωρήσουμε. Υπάρχει μια σειρά ζητημάτων ε, που προέκυψαν από το έγγραφο της διαβούλευσης. Αυτό το στάδιο λοιπόν είναι δύσκολο γιατί δεν μπορούμε να προβλέψουμε ποιο θα είναι το μέλλον αυτών των αρχών. Ε, πώς θα διαρθρώνονται, αν θα έχουν τις ίδιες αρμοδιότητες. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε τώρα είναι να έχουμε μια πολύ στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι το σύστημα υποπτίας θα γίνει πιο ισχυρό μετά από αυτή την αναθεώρηση και θα είναι και ομοιόμορφο ε, στο βαθμό που γίνεται διότι παραμένουν πολλές διακριτικές ευχαίρειες στις διάφορες χώρες που καθιστούν το τρέχον σύστημα μη εναρμονισμένο σε πλήρες ε, επίπεδο. Τώρα, ε, είναι δύσκολη η απάντηση να πω και άλλη μια φορά ότι η τρέχουσα τάση θα παραμείνει, στάση θα παραμείνει μέχρι να δούμε ε, μια αλλαγή στη ροή του πληθωρισμού. Ξέρουμε ότι θέλουμε πληθωρισμό κοντά στο 2% για όλη την Ευρωζώνη, όχι για τη μία χώρα ή την άλλη, που να είναι κάτι ε, που θα παραμείνει, δεν θα συμβαίνει για μία στιγμή. Μπορεί να έχουμε χαμηλό πληθωρισμό, αλλά αυτό είχε να κάνει με την αύξηση των τιμών στον ενεργειακό τομέα. Ε, αν ε, μειωθούν αυτές, μειώνεται και το headline inflation. Έτσι λοιπόν πρέπει να διαρκέσει και να πιστούμε ότι θα διαρκέσει ε, με όλη την νομισματική υποστήριξη που έχουμε ε, χρησιμοποιήσει. Για το τρίτο θέμα που είπατε. Όλοι μας ανησυχούμε, είναι γεγονός. Όλο η οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ενιαίας αγοράς, βασίζεται στο ε, να μοιραζόμαστε τα ωφέλη του ελεύθερου εμπορίου. Βέβαια, αυτά που συνέβησαν τα τελευταία 15-20 χρόνια, στην ουσία μας οδήγησαν στο να έχουμε μεγάλα ωφέλη αλλά και ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν μερίδιο σε αυτά τα ωφέλη από το ελεύθερο εμπόριο και την παγκοσμιοποίηση του ελεύθερου εμπορίου. Πρέπει λοιπόν να βελτιωθούμε σε αυτό το τομέα. Όλοι να έχουν μερίδιο σε αυτά τα ωφέλη. Όλοι όσοι συμμετέχουν στη διαδικασία. Αυτές οι νεοπροστατευτικές όμως στάσεις που ε, αυτή τη στιγμή εκφράζονται τις Ηνωμένε Πολιτείε σίγουρα μας ανησυχούν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πέντρο Σίλβα Περέιρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Ντράγκη, με χαρά μας σας καλωσορίζουμε εδώ. Ας να σας κάνω δύο ερωτήσεις. Η πρώτη έχει να κάνει με την νομισματική πολιτική. Όπως είπατε ξεκάθαρα σήμερα εδώ, οι πιέσει σε εγχώριο επίπεδο, κυρίως από τους μισθούς, δεν μας ε, επιτρέπουν να έχουμε μια διαρκή σύγκληση του πληθωρισμού και βέβαια οι θετικέ τάσεις δεν πρέπει να μας ε, αποτρέπουν από το να παραμένουμε πιστοί στην εστίαση στην ανάγκη για ανάπτυξη. Είπατε ότι χρειαζόμαστε σε μεγάλο βαθμό την νομισματική πολιτική παρόλα αυτά λοιπόν. Να πω λοιπόν ότι ε, αυτό που κατάλαβα είναι ότι δεν έχετε στο άμεσο μέλλον την πρόθεση να σταματήσετε την άσκηση νομισματικής πολιτικής. Το άλλο θέμα έχει να κάνει με την Πορτογαλία. Όπως ξέρετε πρόσφατα η Κομισιόν πρότεινε η Πορτογαλία να βγει από την διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, λαμβάνοντας υπόψη τη μείωση του ελλείμματος και τις θετικές εξελίξεις ε, που έχουν να κάνουν με την οικονομική ανάπτυξη, την μείωση της ανεργίας κτλ. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν ε, να σας ρωτήσω πώς βλέπετε αυτές τις εξελίξεις. Σε αυτό το πλαίσιο η κυβέρνηση της Πορτογαλίας ζήτησε να προκαταβάλει ένα μεγάλο ποσό του δανείου από το δενοτού που έχει λάβει. Θεωρείτε ότι αυτή η καταβολή ενδεχομένως να βοηθούσε στην αντιμετώπιση δυσκολιών σχετικά με τα όρια του προγράμματος εξαγοράς της ε, ΕΚΤ λαμβάνοντας υπόψη βέβαια ότι αυτά τα όρια αυτή τη στιγμή οδηγούν σε μία μείωση των εξαγορών από την ΕΚΤ. Θεωρείτε ότι θα έχετε περισσότερο περιθώριο χειρισμών, να υπάρχουν περισσότερα ομόλογα τα οποία να είναι επιλέξιμα για το πρόγραμμα εξαγοράς της ΕΚΤ. Απάντηση. Για την πρώτη σας ερώτηση η απάντηση είναι ακριβώς η ίδια με αυτή που είπα πριν. Οι εξελίξεις που βλέπουμε στον πληθωρισμό μας δείχνουν ότι η υπερβολική αυτή η επεκτατική η νομισματική πολιτική που έχουμε αυτή τη στιγμή πρέπει να παραμείνει. Οι εξελίξεις ε, στη σύγκληση του, διαδικασία σύγκλησης του πληθωρισμού πρέπει να μας καταδείξουν ότι η κατάσταση θα μας οδηγήσει στους στόχους μας, ε, θα είναι αυτό και θα παραμείνει. Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε το επόμενο Συμβούλιο Νομισματικής ε, Πολιτικής και τις νέες προβλέψεις ε, για το προσωπικό που θα μας δώσουν και νέες πληροφορίες για το θέμα αυτό. Στο δεύτερο ερώτημά σας να απαντήσω ότι όντως έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος στην Πορτογαλία σε όλα τα επίπεδα και αυτό είναι το πρώτο σημείο που θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Δεύτερον, εν τούτης, υπάρχουν πολλά σημεία που παραμένουν τροτά, ειδικά στον τραπεζικό τομέα, που έχουμε μεγάλο αριθμό MPLs, ε, όπως ε, και σε άλλες χώρες της περιφέρειας και πρέπει αυτά τα τροτά σημεία να τα αντιμετωπίσουμε πρώτον για τη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος αλλά και για να εκμεταλλευτούμε πλήρως τη δυνατότητα των πορτογαλικών τραπεζών να υποστηρίξουν και να χρηματοδοτήσουν την πραγματική οικονομία. Τα MPL είναι ε, ένα βαρύδι ε, προς ε, την παροχή πιστώσεων. Το τρίτο θέμα που θέσατε έχει ως απάντηση ότι δεν το νομίζω. Δεν νομίζω ότι έχει σχέση η προκαταβολή αυτού του δανείου με τα όρια της ποσοτικής χαλάρωσης. Ευχαριστώ. Κύριε Λάγκεν. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, που έρχεστε τακτικά να μας δείτε. Έχω τρεις διαφορετικές ερωτήσεις. Η μία έχει να κάνει με την κίνηση του ρευστού χρήματος και το τεράστιο κενό φόρου προσθέμενης αξίας, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες που μας λένε ότι όπου είναι πολύ μεγάλο το κενό στο φόρο προσθέμενης αξίας, είναι και μεγάλη κυκλοφορία του ρευστού. Με την κατάρριξη των, ε, των χαρτογράφων του, των 500, των 500 ευρώ και αντίστοιχα των ε, μικρών ε, νομισμάτων των 5 cents. Αυτό ήταν το ένα. Το άλλο ήταν το Euro Clearing που ανέφερε και ο συνάδελφος νωρίτερα και σε συνδυασμό με το Brexit. Θεωρείτε ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια μορφή συνεργασίας με το Λονδίνο στηριζόμενη στην, στο σύστημα που έχει τώρα η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών και πιστεύετε ότι θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών να αναλάβει το ρόλο της στο πλαίσιο της ΕΚΤ. Και η άλλη, η τρίτη ερώτηση, έχει να κάνει με την νομοθεσία των ΗΠΑ, γιατί χρειάστηκαν χρόνια μέχρι ότου να υλοποιηθεί το Frank Act. Είχε ξεκινήσει με τη, η συζήτηση με τον ε, Bush, με τον Ομπάμα μετά, μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι μας επιφυλάσσουν οι ΗΠΑ με τις προτάσεις του νέου εκλεγέντος Προέδρου. Πάντως ε, λέει ότι θέλει να, θέσει, θέλει να ακυρώσει τον νόμο Dodd Frank και γι' αυτό να ρωτήσουμε, θέλω να ρωτήσω εάν βλέπετε πράγματι τους κινδύνους ή αν η κατάσταση στην πραγματικότητα παρουσιάζει διαφορετική εικόνα. Ευχαριστώ. Απάντηση για την πρώτη σας ερώτηση. Εάν η εκτεταμένη χρήση ρευστού μπορεί να σχετίζεται με φοροδιαφυγή και δίφρο φόρου προσθεμένης αξίας. Είναι πιθανό κάτι τέτοιο να συμβαίνει. Και σε αυτή τη χρονική στιγμή δεν έχω να διαθέσω συγκεκριμένα στοιχεία. Πολύ ευχαριστώ να σας απαντήσω γραπτός. Είναι πολύ πιθανό όμως να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Δεύτερον, για την διεθνή συνεργασία. Είναι βεβαίω θεμελιώδη για την καταπολέμηση τη φοροδιαφυγή, είτε πρόκειται για τη χρήση ρευστού χρήματο, είτε με άλλη μορφή. Είναι αναμφίβολη η συμφωνία όλων των κυβερνήσεων ουσιαστικά στο θέμα αυτό και ανεξαρτήτως τι θα συμβεί, και βεβαίω ξέρετε ποια είναι η πεποίθησή μου, όσο λάθο και αν μπορεί να τη θεωρήσετε. Εγώ πιστεύω ότι με τι διαπραγματεύσει στο όνομα Βασίλειο, με, το, με την Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή, η συνεργασία για την καταπολέμηση φοροαποφυγής, φοροδιαφυγής θα πρέπει να διατηρηθεί, θα διατηρηθεί. Είναι κάτι το οποίο έχουν επαναλάβει όλες οι χώρες και στην πρόσθετη πρόσφατη συνεδρία των Υπουργών των Οικονομικών στο G7, στο πλαίσιο του G7, υπάρχει σχετική αναφορά και μάλιστα και σχετική φράση στο τελικό ανακοινωθέν τύπου. Δεύτερη ερώτηση για την ε, Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών και την ΕΚΤ. Δεν είναι απαραίτητο να συμβεί αυτό, γιατί έχουν διαφορετικές λειτουργίες η αρχή τραπεζών, είναι ρυθμιστική αρχή, η ΕΚΤ ε, είναι λίγο πολύ αρχή εποπτείας και έτσι βεβαίως δεν είναι δική μας δουλειά γιατί εσείς θα αποφασίσετε ως νομοθέτες. Πιστεύουμε ότι οι δύο αρχές θα πρέπει να παραμείνουν σε λειτουργία παράλληλα γιατί ε, απευθύνονται και σε διαφορετικές τράπεζες, σε διαφορετικές χώρες. η γεωγραφική περίμετρος δηλαδή δραστηριοποίηση είναι διαφορετική. Η τελευταία σας ερώτηση είχε να κάνει ναι. Είναι νομίζω πρόωρο. Να πούμε αν η αναθεώρηση της χρηματοοικονομικής χρηματοπιστικής νομοθεσίας από πλευράς της κυβέρνησης των ΗΠΑ μπορεί να οδηγήσει σε τροποποιήσεις στο τμήμα αυτό της νομοθεσίας που αφορά την ρευστοποίηση και το ενεργητικό των τραπεζών. Ή το τμήμα αυτό που έχει να κάνει περισσότερο με τη ρύθμιση της αγοράς. Καρόνες Βόλκερε, παραδείγματι, market making και άλλα σχετικά θέματα που έχουν να κάνουν περισσότερο με την ε, νομοθεσία ρύθμιση αγοράς. Ή εάν θα καλύψει και τα δύο αυτή η εξέλιξη. Είμαστε σε μια διαρκή επικοινωνία. Αυτή τη στιγμή όμως ακόμη δεν έχουμε σε φυγικό. Αυτό που επισημαίνετε και εσείς έχει πολύ μεγάλη σημασία γιατί αναλόγως ότι μπορεί να αποφασιστεί. Εμείς θέλουμε και ελπίζουμε μια παγκόσμια ε, συμφωνία στα θέματα των ε, προϋποθέσεων, των προδιαγραφών για κεφαλαιοκική ευστότητα για να λειτουργήσει σωστά το σύστημα. Ευχαριστώ Μόργανο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε. Κύριε Ντράκη. Είναι γνωστό ότι καθήκον της ΕΚΤ είναι η σταθερότητα σε ΕΚΤ και όχι μόνο βέβαια, όχι ιδιαίτερος υποστήριξη της απασχόλησης, αλλά είναι γνωστό ότι χωρίς αύξηση της απασχόλησης, χωρίς μια καλή απασχόληση, ε, η δυναμική της ε, ανάπτυξης και του πληθωρισμού θα παρέμενε μάλλον αρνητική, όπως άλλωστε και εσείς τους τελευταίους μήνες έχετε επανειλημμένως υπογραμμίσει. Θα θυμάστε ασφαλώς ότι πρόκειται γιατί, γιατί το έχετε πείτε στη Φραγκφούρτη, είτε εδώ, στην Επιτροπή μας, ότι μια νομισματική πολιτική δεν μπορεί να είναι ο μοναδικός μηχανισμός ενίσχυσης και υποστήριξης της ανάπτυξης στην Ευρωζώνη και ότι χρειάζονται μέτρα κατάλληλα ε, και φορολογική πολιτική. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα και δημοσιονομική πολιτική, Γι' αυτό θα ήθελα λοιπόν να διατυπώσω τα εξή ερωτήματα. Πιστεύετε ότι η νομισματική πολιτική θα ήταν πιο αποτελεσματική και ω προ την διαμόρφωση, εάν υπήρχε μια διαμόρφωση των δημοσίων δαπανών που να ευνοεί την ανάπτυξη με μια φορολογική πολιτική συντονισμένη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επεκτατική όπω αυτό που είχε πει ο κύριο Μοσκοβίση το Δεκέμβριο του 2016. Δεύτερη ερώτηση. Πιστεύετε ότι η δημοσιονομική πολιτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα μπορούσε να έχει ένα κατάλληλο policy mix με μία δημοσιονομική δυναμική της Ευρωζώνης που θα χρηματοδοτούνταν από τους ιδίους πόρους και αν υπήρχε αυτή η δυνατότητα για ιδίους πόρους για τη χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωζώνης τι είδους μεγέθη θα έπρεπε να διαθέτει αυτός ο ευρωπαϊκός προπολογισμό για να αντισταθμίσει τους οικονομικούς κύκλους. Ναι, έχω πει πολλές φορές ότι η νομισματική πολιτική θα μπορούσε να είναι πολύ πιο αποτελεσματική εφόσον υπάρχουν πολιτικές δημοσιονομικές, διαθροτικές πολιτικές που έρχονται να αυξήσουν τις ε, ε, δυνατότητες ανάπτυξης. Οι δυνατότητες που έχει αυτή τη στιγμή με βάση την παρούσα δημοσιονομική πολιτική η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ε, είναι ότι εμείς πρέπει να έχουμε μια, ένα ουδέτερο δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Και αυτό είναι το σωστό. Αυτή είναι η αξιολόγησή μας τουλάχιστον ως ΕΚΤ. Θεωρούμε ότι η παρούσα ουδέτερη δημοσιονομική προσέγγιση είναι η κατάλληλη ε, σε ό,τι αφορά το ποιο είναι το κατάλληλο μείγμα πολιτικής, έτσι. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο ερώτημά σα τώρα. Εγώ νωρίτερα αναφέρθηκα στον ευάλωτο χαρακτήρα, στον έστραυστο χαρακτήρα της Νομισματικής Ένωσης επειδή δεν έχει ολοκληρωθεί η Ένωση. Μέρος αυτού που μένει να γίνει για να ολοκληρωθεί είναι ότι δεν έχουμε μια δημοσιονομική δυνατότητα. Είναι μια έννοια η οποία είναι βασική για κάθε νομισματική ένωση και για κάθε ε, νομισματική αρχή ή θεσμικό όργανο. Πώ όμω θα φτάσουμε στη δημιουργία αυτή τη νομισματική δυνατότητα, Ποια είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν. Έχω πει πολλές φορές δεν ξέρω αν το είπα και εδώ, ότι χρειαζόμαστε δύο πυλώνες για τη δημιουργία αυτής τη δημοσιονομική δυνατότητας. Το ένα πυλώνας είναι η εμπιστοσύνη και ο άλλο είναι η σύγκληση. Η εμπιστοσύνη έχει να κάνει με το ότι για να έχουμε μια κοινή δημοσιονομική δυνατότητα με κοινέ εξουσίε πρέπει να εμπιστευόμαστε εμέν του δε. Πρέπει να πιστέψουμε ότι δεν μπορούν να είναι κάποιοι μόνιμα πιστωτές και κάποιοι μόνιμα οφειλέτες. Δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε μια μόνιμη μεταφορά ε, κεφαλαίων προς την διακατεύθυνση. Πρέπει να υπάρχει αυτή η ένωση για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα σοκ, της αστάθειες, για να μπορούμε να παραλύθουμε σαν σημείο ισορροπίας. Το δεύτερο όμω που είναι ακόμα πιο σημαντικό είναι ότι οι χώρε που συμμετέχουν σε μια νομισματική ένωση δεν μπορεί να είναι πολύ ετερογενείς μεταξύ του. Πρέπει να συγκλίνουν. Και η σύγκληση σημαίνει διαθροτικές μεταρρυθμίσεις. Και οι διαθροτικές μεταρρυθμίσεις δεν είναι ίδιες σε όλες τι χώρες. Η κάθε χώρα τη νομισματικής Ένωση χρειάζεται ε, συγκεκριμένες διαθροτικές μεταρρυθμίσεις, διαφορετικές. Είναι δύσκολο λοιπόν να θεσπίσουμε ένα κατάλογο που να είναι σωστό για όλου. Σίγουρα πάντω πρέπει να υπάρχει σύγκληση. Σύγκληση προ τα πού. Σύγκληση προ υψηλότερου ρυθμού ανάπτυξη. Από κοινού. Αρχίζουμε να το βλέπουμε κάπω αυτό. Βλέπουμε ότι η ανάπτυξη σε προσθέμενη αξία ε, είναι πολύ λιγότερο ε, άνηση από ό,τι πριν την κρίση. Ευχαριστώ. Ναι, ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ, κύριε Δράκη, που εδώ. Οι πληρωμές στο, της μετρητής είναι ένα από, το πιο, από τα πιο συνηθισμένα μέσα που χρησιμοποιεί το οργανωμένο έγκλημα, οι μαφιόζικε οργανώσεις, η φοροαποφυγή. η Ινδία λοιπόν το προηγούμενο Νοέμβριο προχώρησε σε μια νομοθέτηση που σκόχο έχει ακριβώς ε, να καταπολεμήσει αυτή η φοροαποφυγή και το μαύρο χρήμα που κυκλοφορεί καταργώντας λίγο πολύ τις πληρωμές της μετρητής και αυτό έχει ενισχύσει ιδιαίτερα την οικονομία της χώρας. Στην Ιταλία, δυστυχώς, είναι ακόμη πολύ συνηθισμένη η χρήση των μετρητών και λόγω του υψηλού κόστους φερειπίν τη συνδρομή σε μια πιστοτική κάρτα με 3,6% ε, για τον έμπορο συνδρομή και 35 ευρώ περίπου για τον καταναλωτή ε, κατά μέσο όρο. Είχε γίνει λοιπόν πρόταση από την Ιταλική Οργάνωση Τραπεζών η πιστοτική κάρτα να χρησιμοποιείται ιδιαιτέρως σε θέματα ε, κατάρτισης των φορολογικών δηλώσεων και των φορολογικών ελέγχων. Μπορεί δηλαδή η Ιταλία να ξεκινήσει μια πολιτική ενίσχυση της χρήσης του πλαστικού χρήματος, ξέροντας βέβαια ότι μια τέτοια πολιτική θα σήμαινε ταυτόχρονα και την μείωση της χρήσης των μετρητών. Επομένως, ε, θα περιόριζε το πεδίο για τις παράνομες δραστηριότητες. Και άλλη μια ερώτηση Η Ιταλία ξεκινάει ένα σύστημα που θεωρείται από τους οικονομικούς παράγοντες μάλλον επικίνδυνο, ότι δηλαδή όλες οι ε, χρηματοπιστωτικές συναλλαγές που γίνονται online μπορεί να οδηγήσουν σε μία πρόβλεψη ότι θα είναι αρνητικές εξελίξεις των χρηματιστηρίων. Ε, μια, ένα θεματολόγιο δηλαδή το οποίο ενισχύεται από την προοπτική για πρόορε εκλογέ και θα μπορούσε να οδηγήσει σε ακόμη χειρότερα προβλήματα για την οικονομία τη χώρα. Μήπω θα έπρεπε λοιπόν να έχουμε μια διαφορετική πολιτική και να μην γίνουν πρόορε εκλογές για να ενισχυθεί η τελική οικονομία. Κύριο Δράγκη, για τη δεύτερη ερώτηση, συγγνώμη, αλλά δεν έχω ιδιαίτερες, ε, ιδιαίτερα σχόλια να κάνω. Δημοκρατία έχουμε, εκλογέ προβλέπονται πάντα. Δεν μπορεί κανεί να διατυπώσει κρίση και πάντως θα είμαι εγώ αυτό ο οποίο θα κάνει μια τέτοια κρίση για το πότε θα πρέπει να γίνουν οι εκλογέ στα αγγλικά. Το άλλο ερώτημα έχει να κάνει με τη χρήση των ρευστών, του, των μετρητών και το συσχετισμό τους με τις εγκληματικέ δραστηριότητες. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι και μάλιστα η ΕΚΤ έχει αναλάβει δράση παρελειμμένο στο πεδίο αυτό με τη σταδιακή μείωση μέχρι και εκμηδενισμό της παραγωγής εν τέλει των χαρτονομισμάτων των 500 ευρώ για τα επόμενα χρόνια που σχεδιάζεται. Πρέπει όμως και να αναγνωρίσουμε το γεγονός ότι υπάρχουν διαφορετικές προτιμήσεις σε κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάθε λαός έχει διαφορετικές προτιμήσεις προς τη χρήση των μετρητών. Και ταυτόχρονα, όντως, τα μετρητά χρησιμοποιούνται, αξιοποιούνται για δραστηριότητες όχι νόμιμες, που μπορεί να είναι και ποικίλε. Πρέπει λοιπόν να επαγρυπνούμε και να δραστηριοποιούμαστε. Βεβαίως να γνωρίζουμε τη σημασία της χρήσης του αιών ρευστών, που πολλές χώρες έχουν υποστηρίξει και πολλοί λαοί εκφράζουν σε διάφορες χώρες της Ευρωζώνης. Ε, ίσως θα ήταν περισσότερο να κοιτάξουμε να μην υποστηρίζει χρήση των ρευστών τι εγκληματικέ δραστηριότητε. Αυτό πρέπει να ελέγξουμε. Μιλήσατε για την δυνατότητα, η πιστοτική κάρτα Φερρυπίν, να χρησιμοποιείται για τις φορολογικές δηλώσεις. Γιατί όχι. Οι εθνικές αρχές όμως έχουν μεγάλο περιθώριο επιλογών και χειρισμών για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και για την αξιολόγηση και τον περιορισμό αυτής. Είτε πρόκειται για χρήση μετρητών είτε όχι και βεβαίως οι εθνικές αρχές και φορείς δραστηριοποιούνται, αντίστοιχα δραστηριοποιούνται βέβαια και οι φορείς σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Λίνα Τζιλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δύο σημεία. Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι η ανεργία στην Ευρωζώνη είναι η χαμηλότερη τα τελευταία 8 χρόνια. Όμω μέρος τη επιτυχία αυτή έχει να κάνει με το quantitative easing ε, τη ε, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Είπατε σήμερα ταυτόχρονα ότι χρειαζόμαστε υψηλότερη παραγωγικότητα υψηλότερη ανάπτυξη και αυτό χρειάζεται καινοτομία. Η καινοτομία στον χρηματοοικονομικό τομέα είναι ένα σημείο κλειδί, αλλά και σε άλλου τομεί. Μόλι το G7 ε, συζητήθηκε το θέμα τη κλιματική αλλαγή. Ο κύριος Τραμπ αρνείται βεβαίω να ακολουθήσει για την ώρα. Εάν δούμε όμω τι έγινε στο COP21 στο Παρίσι, η Συμφωνία για την Αλλαγή του κλίματο, όπου συμφωνή, που συμφωνήθηκε από τους G20, έχει να κάνει με ένα σαφέ στρατηγικό μήνυμα για να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην πράσινη χρηματοδότηση. Τώρα αναγνωρίζω ότι είναι σημαντικό αυτό που είπατε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα, δηλαδή να είναι ουδέτερη, να υπάρχει ουδετερότητα, αλλά υπάρχει σαφή δέσμευση από την Ευρώπη να βελτιώσουμε την ποιότητα του περιβάλλοντος μας. Μήπως ήρθε η ώρα για τα 60 δις που ε, επενδύει κάθε μήνα η Ευρωπαϊκή Ενταγή Τράπεζα για το quantitative easing ε, να ακολουθεί μια πιο ε, διαφανή διαδικασία σε ό,τι φέρα το QE και τα χρήματα αυτά να πηγαίνουν και σε πιο πράσινες δραστηριότητε. Το δεύτερο ερώτημά μου τώρα αφορά τις CCPs. Απαντήσατε προηγουμένω στον συνάδελφο των Von Βάιτ και είπατε ότι θα συνεχίσετε το παρόν καθεστώς και τα παρόντα εργαλεία για να, καταπο... να αντιμετωπιστούν τα συστημικό κίνδυνο CCPs από τρίτες χώρες. Τι αναμένετε ε, από τη συνεργασία με την Τράπεζα της Αγγλίας και πώς αξιολογείτε τα επιχειρήματα αυτών που είναι κατά μιας ε, ε, πολιτικής Eurolocation που λέγοντα ότι αυτό θα αυξήσει ε, το τραπεζικό κεφάλαιο. Thank you. Um, on your first question... Ναι, για το πρώτο σας ερώτημα. Εμείς όταν σχεδιάσαμε το πρόγραμμα ε, αγοράς ε, ομολόγων για τις επιχειρήσεις. Αυτό το πρόγραμμα εμείς είχαμε κατά νου ε, ζητήματα νομισματικής πολιτικής, ζητήματα διαχείρισης κινδύνου και βεβαίως ίσως, ίσο ανταγωνισμό, ίσες ευκαιρίες. Αυτό απαντάει <laughs> λίγο και στο ερώτημα που τέθηκε νωρίτερα κατά πόσο ε, κάποιες, <laughs> κάποιες επιχειρήσεις ε, θα λύνουν περισσότερο από ό,τι άλλες. Όχι. Η απάντηση είναι όχι. Είχαμε πει ότι το κριτήριο είναι το level playing field, δηλαδή ίσες ευκαιρίες, ίσο πεδίο ευκαιριών για όλους. Τώρα από εκεί και πέρα, τα κριτήρια επιλεξιμότητας είναι αρκετά διευρυμένα, έτσι ώστε πολλές πράσινες εταιρείες και βεβαίως τα ομόλογά τους να μπορούν να αγοραστούν από, το, πρόγραμμα τα προγράμματά μας. Η απάντηση στο ερώτημά σας λοιπόν είναι ε, ότι εσείς θέλετε ένα πρόγραμμα που να, ε, ε να απευθύνεται αποκλειστικά ε, στην πράσινη ανάπτυξη. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Τώρα, το πρόγραμμά μας δίνει τη δυνατότητα σε εταιρείε που πάνε προς την πράσινη χρηματοδότηση να συμμετάσχουν. Η απάντηση είναι ναι. Το δεύτερο ερώτημά σας τώρα. Η παρούσα κατάσταση. Αναφερθήκατε σε δύο ζητήματα, τα CCPs και οι τράπεζες και τι θα γίνει με την μετεγκατάσταση τραπεζών. Τι θα, πού θα οδηγήσει αυτό. Ε, βεβαίως, η πρόσφατη απόφαση του Εμένου Βασιλείου να φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργεί ανησυχίες ό,τι φοράει τι δυνατότητε του Ευρωσυστήματος να ελέγξει τις επιπτώσεις των αρχών ε, offshore clearing ε, και ταυτόχρονα στα, να παραμείνει σταθερότητα του ευρώ. Ε, εμείς καλωσορίζουμε το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να εξασφαλίσουμε την υγιή, ε, την υγεία, αν θέλετε, των ε, CCP που είναι συστημική σημασία. Στις 4 Μαΐου στην θετική ανακοίνωση αναφέρθηκαν μια σειρά από δυνατότητε ενισχυμένη εποπτεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ε, προϋποθέσεις relocation μετεγκατάστασης. Είναι κάπως νωρίς βεβαίως για να σχολιάσουμε το πλαίσιο αυτό, διότι δεν έχει εκριθεί ακόμα. Πάντως τα, οι αυξημένες απαιτήσει κεφαλαϊκές που αναφέρεται ως κίνδυνο είναι σημαντικές κυρίως για τις τράπεζες και όχι για τις CCPs, αλλά μπορεί να αποδειχθούν σημαντικές και για τα CCPs. Σαφώς. Θα πρέπει να το εξετάσουμε προσεκτικά και θα πρέπει βεβαίως να ακούσουμε κιόλας, να πάνε η χώρα μια διαβούλευση και με τον κλάδο. Εμείς δεν συμμετέχουμε στη διαπραγματευτική, έτσι. Ε, είμαστε ρεθυμένοι να δώσουμε τη συμβουλή μας να μας ζητηθεί, αλλά δεν συμμετέχουμε επισήμως σε αυτή τη διαπραγμάτευση. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ. Ο κύριος Νίναρχοκμα. Χόκμαν. Ευχαριστώ. Πάντοτε με εντυπωσιάσει πόσο πολύ θέλετε εδώ στο σώμα μας και στο δικό σας να συζητάτε τις θεσμικές αλλαγές και όχι τις δύσκολες πολιτικές αποφάσεις που χρειάζονται για τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις σε επίπεδο ευρωπαϊκό και σε επίπεδο κράτους μέλους. Νομίζω κάποιες φορές είναι σαν να ψάχνεις να βρεις τα κλειδιά ε, το φως του δρόμου αντί να ψάχνεις να βρεις που τα ε, μιλάμε για την νομισματική πολιτική και την ανάπτυξη, αντί να μιλάμε για την έλλειψη ανάπτυξης. Όπως αναφέρατε πριν, υπάρχουν διάφορα επίπεδα ανάπτυξης στα κράτη-μέλη. Οι προϋποθέσεις για την νομισματική πολιτική διαφέρουν. Ταυτόχρονα όμως και τα επίπεδα δυνητικής ανάπτυξης και αντιμετώπισης ε, του χάσματος σε επίπεδο παραγωγής είναι ε, μεγάλο ζήτημα. Το παράδειξο είναι ότι οι χώρες που χρειάζονται την περισσότερη ανάπτυξη έχουν, διατρέχουν τον κίνδυνο να έχουν προβλήματα λόγω του πληθωρισμού και των ε, επιτοκίων πριν έρθει το υψηλό ποσοστό ανάπτυξης. Το ερώτημά μου θα είναι δύσκολο να το απαντήσετε, όμως είναι πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Να την πάω και ένα βήμα παραπέρα την ερώτησή μου. Δεν θα έπρεπε κατά κάποιο τρόπο να θέσουμε στόχους στα διάφορα κράτη-μέλη για το επίπεδο δυνητικής ανάπτυξης για να μπορέσουμε να μετρήσουμε και το μέγεθος των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που χρειάζονται, γιατί όταν είναι μικρή ανάπτυξη έχουμε μεγάλη ανάγκη για τέτοιες μεταρρυθμίσεις. Απάντηση. Συμφωνώ με αυτά που είπατε. Η ετερογένεια. Υπό την έννοια δηλαδή Ε, διαφορετικών δυνατοτήτων ανάπτυξης, ε, αν όχι δραματικά διαφορετικών ε, δυνατοτήτων ανάπτυξης, είναι μία από τις αδυναμίες στην Νομισματική Ένωση. Και η απάντηση είναι μία και μοναδική, να γίνουν οι απαραίτητες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Τώρα, τι θα μπορούσε να κάνει ένα κοινό πλαίσιο για να βοηθήσει μια τέτοια διαδικασία. Υπό μία έννοια έχουμε Τώρα στα σπάργανα με το, ε, ε, με το CSR και το οικονομικό εξάμεινο, της στάση δηλαδή ένα χώρα έχουμε στα σπάργανα ένα τέτοιο κοινό πλαίσιο. Η απάντηση λοιπόν είναι ότι πρέπει να ενισχύσουμε σημαντικά αυτό το κοινό πλαίσιο. Πρέπει να δημιουργήσουμε κάτι που εσείς ήδη προτείνατε, ένα σύστημα συγκρίσιμων όρων, ένα benchmarking, ε, όπου οι χώρες ε, θα κάνουν, όπως κάνουν και με τις δημοσιονομικές τους πολιτικές, μια σύγκριση των μεταρρυθμίσεών τους και η πρόοδος θα συζητείται από κοινού μεταξύ των κρατών μελών. Αυτή είναι η απάντηση σε αυτή την τρέχουσα συγκυρία νομίζω. Μια επερώτηση να κάνω διότι πλήρως συμφωνώ μαζί σας, όμως κατά κάποιο τρόπο θεωρώ ότι από τη στιγμή που μιλάμε για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, μιλάμε για ωραία λόγια, για... είμαστε απλώς ευγενικοί. Λέμε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Από την άλλη, ξέρουμε πολύ καλά ποιες είναι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται, αλλά πολιτικά είναι ευαίσθητο το ζήτημα είμαστε αυστηροί ως προς το σύμφωνο σταθερότητας. Ε, όχι τόσο, αλλά τέλος πάντων πρέπει τυπικά να είμαστε αυστηροί. Από την άλλη είμαστε ιδιαίτερα ασαφείς όσον αφορά τους πιο ε, βασικούς ε, παράγοντες ε, σταθερότητας και ανάπτυξης. Απάντηση. Φυσικά. Και ένας τρόπος για να το ξεπεράσουμε αυτό είναι από τη μία να ενισχύσουμε το ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διότι αυτή είναι ο θεματοφύλακας των συνθήκων του ε, Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και μπορεί να γίνει, αν όχι ο θεματοφύλακας, σίγουρα ο βασικός παίκτη που θα διασφαλίσει ότι οι χώρες σέβονται αυτή τη διαδικασία του benchmarking που ε, στην ουσία δείχνει την πρόοδό τους ε, στις ε, ε, μεταρρυθμίσεις και απ' την άλλη θα πρέπει να ενισχύσουμε το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και τις συστάσεις αναχώρα διότι αυτό που θέλουμε να ξεπεράσουμε είναι να μην είναι απλώς εθνικό ζήτημα οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, διότι δεν είναι πλέον εσωτερικό ζήτημα είναι η ετερογένεια που δημιουργεί την ε, αυτή κατάσταση στην νομισματική ένωση. Ο κύριος Μαριάς. Ε, επανέρχομαι στο θέμα της Τράπεζας της Ελλάδος που σας ανέφερα προηγουμένως. Διότι η Ελλάδα είναι εκτός ποσοτικής χαλάρωσης, το ξέρουμε και μάλιστα... Should I start from the beginning? You don't have interpretation in Greek? Is it Κύριε Πρόεδρε, επανέρχομαι στο θέμα της Τράπεζας της Ελλάδος, διότι η Ελλάδα ως χώρα είναι εκτός ποσοτικής χαλάρωσης και μάλιστα εσείς, απαντώντας πριν λίγο σε μένα, βάλατε και νέους σκληρούς όρους προκειμένου να μπει η Ελλάδα στο QE, αλλά η Τράπεζα της Ελλάδος συμμετέχει στο QE και έχει δαπανίσει 42,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Και τη στιγμή αυτή ξέρουμε ότι αγόρασε ομόλογα διεθνών οργανισμών όπως μου απαντήσατε, αγόρασε ορμόλογα του ESM και του EFSF. Δηλαδή αγόρασε ομόλογα των δανειστών οι οποίοι μας δανείσαν και μας επέβαλαν μνημόνιο. Λοιπόν, η ερώτηση που σας έκανα είναι συγκεκριμένη. Μπορούσε η Τράπεζα της Ελλάδος να αγοράσει ομόλογα ελληνικών επιχειρήσεων και ελληνικών τραπεζών. Διότι το σύστημα CBPP3 είναι τελείως διαφορετικό από το PSPP Δηλαδή είναι άλλο πράγμα να αγοράζεις κρατικά ομόλογα, τα οποία βάλατε περιορισμούς, και άλλο να αγοράζεις ομόλογα ελληνικών εταιριών. Για ποιο λόγο κάνατε αυτό το διαχωρισμό. Και δεύτερον, στο θέμα της πρότασης που σας έκανα προηγουμένως και αναδεικνύεται από τη συζήτηση που υπάρχει, υπάρχει ετερογένεια μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλες χώρες είναι σε ανάπτυξη, λέω ότι στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει ετερογένεια. Άλλες χώρες είναι σε ανάπτυξη, άλλες είναι σε ύφεση. Εσείς εφαρμόζετε μια ενιαία νομισματική πολιτική. Εγώ δεν είπα να την αλλάξετε αυτή. Εγώ είπα να την εφαρμόσετε. Όμως να δώσετε την ευκαιρία σε κάθε εθνική κεντρική τράπεζα να εφαρμόσει τη δική της νομισματική πολιτική για την δικιά της οικονομία χρησιμοποιώντας QE. I'm going to, to seconds χρησιμοποιώντας QE στο ύψος που έχει ποσοστό μέσα στο κεφάλαιο της Κεντρικής Τράπεζας. Δηλαδή, η Ελλάδα... Την ίδια ερώτηση, απάντηση, ερώτηση με πριν κάνατε. Δεν κατάλαβε την ερώτηση και δεν απάντησε. Είναι η τρίτη φορά που κάνετε αυτή την ερώτηση. Τώρα έχει περισσότερο χρόνο για να απαντήσει ο κύριος Δράγκη όμως. Νομίζω ότι απάντησε αυτή την ερώτηση πριν. Για το πρώτο θέμα που θέσατε, το κάθε QE έχει τα δικά του κριτήρια επιλεξιμότητας. Τα ομόλογα των τραπεζών δεν είναι μέρος του προγράμματος της ποσοτικής χαλάρωσης σε καμία χώρα. Οπότε αυτό εξαιρείται. Τα εταιρικά ομόλογα όμως είναι στο σύστημα. Ναι, όταν και αν μπει η Ελλάδα στο πρόγραμμα, θα δούμε τότε τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Ευχαριστώ. Πρέπει εδώ να ολοκληρώσουμε. Ζητώ συγγνώμη που δεν έχουμε χρόνο για το Catch the Eye, αλλά έχει κλείσει αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης, ο νομισματικός διάλογος με τον κύριο Μάριο Ντράγκη ως πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και περνάμε στη δημόσια ακρόαση με τον Μάριο Ντράγκη ως Πρόεδρο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα δύο λεπτών και μετά θα γίνει η δημόσια ακρόαση με τον κύριο Ντράγκη ως πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου. Έχουμε δυστυχώς λίγο χρόνο στη διάθεσή μας. Απροσδόκητα. Λοιπόν, είμαστε εδώ το σημείο 3 της ημερήσιας διάταξης που είναι η δημόσια ακρόαση με τον Μάριο Τράγκη ως πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου. Για να μην χάνουμε χρόνο δίνω αμέσως το λόγο στον κύριο Τράγκη. Ευχαριστώ. Αγαπηξιότιμα μέλη της ε, Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων. Με χαρά μου βρίσκομαι σήμερα ως Πρόεδρος ε, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου. Ο μοναδικός ε, ρόλος και η οπτική γωνία του Συμβουλίου σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε όλους τους τομείς, μας επιτρέπει να ταυτοποιήσουμε και να, τους κινδύνους και να προσπαθήσουμε να τους μετριάσουμε. Αυτούς δηλαδή τους κινδύνους που προέρχονται από τις αλλαγές στη δομή του χρηματοπιστωτικού συστήματος, οι οποίες μας δίνουν πολλές δυνατότητες να χρηματοδοτήσουμε την πραγματική οικονομία, αλλά καθώς υπάρχει διαμεσολάβηση στο χρηματοπιστωτικό τομέα, η οποία περνάει από τις τράπεζες στις μη τράπεζες, πρέπει να βρούμε τα τροτά σημεία. Θα πρέπει να δούμε και ποια θα είναι τα εργαλεία που θα μας βοηθήσουν να μειώσουμε τους κινδύνους στην σταθερότητα, τη χρηματοπιστωτική, ανεξάρτητα του που αυτή εμφανίζεται. Η μακροπροληπτική πολιτική μας βοηθά σε αυτό, να δημιουργήσουμε ένα ανθεκτικό σύστημα. Γι' αυτό θα ήθελα να μιλήσω για τη δουλειά που κάνει το Συμβούλιο σε αυτό το σημείο. Θα σας μιλήσω λοιπόν για την εποπτεία των μη τραπεζικών πιστοτικών δραστηριοτήτων. Έχουμε το δεύτερο EU Shadow Banking Monitor. Είναι μια έκθεση η οποία αποτελεί βασικό στοιχείο του πλαισίου που έχει το Συμβούλιο για τους κινδύνους ε, και μας δίνει μια γενική εικόνα για τις δραστηριότητες. Για παράδειγμα, το συνολικό σύστημα μη τραπεζικών πιστοτικών δραστηριοτήτων ε, που ε, περιλαμβάνει δηλαδή όλες τις οντότητες ε, εκτός από τις τράπεζες, τα ασφαλιστικά και τα συνταξιδοτικά ταμεία, π.χ. αμοιβαία κεφάλαια βραχυπρόθεσμων επενδύσεων, εκπροσωπεί σήμερα το 38% των συνολικών κεφαλαίων του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού τομέα όπως αυτός ε, ε, αποτυπωνόταν στα τέλη του 2016. Παρόλο που η ανάπτυξη σε αυτόν τον τομέα μειώθηκε το 2016, από το 2012 έχει αυξηθεί κατά 30%. Υπάρχουν διασυνδέσεις λοιπόν με άλλους, ε, άλλα σημεία του χρηματοπιστωτικού τομέα που είναι σημαντικές. Γι' αυτό οι μακροπροληπτικές αρχές πρέπει να προσέχουν για να δουν ποιοι είναι οι κίνδυνοι και τα τροτά σημεία που αναδύονται. Το EU Shadow Banking Monitor τονίζει ακριβώς αυτούς τους κινδύνους, ρευστότητα, μόχλευση, διασυνδεσιμότητα, ε, είναι βασικά θέματα που συζητούνται σε αυτή την έκθεση. Θα ξεκινήσω με τον κίνδυνο για την ρευστότητα και για τη μόχλευση που σχετίζεται με διάφορα επενδυτικά ε, κεφάλαια. Μιλάω, ας πούμε, για εξαγοράσιμες ε, εποχές, οι, ε, μετοχές η σε ημερήσια επίπεδο, οι οποίες ε, την χάνουν ιδιαίτερης ε, μόχλευσης, η οποία η από την πλευρά της μπορεί να δημιουργήσει πιέσεις στο σύστημα και να οδηγήσει σε έκτακτες πωλήσει, αυτές τις fire, λεγόμενες fire sales. Και έχουμε τελικά μία κίνηση των τιμών, ε, έλλειψη ρευστότητας ε, ε, και μία διασυνδεσιμότητα με τη μόχλευση. Έτσι λοιπόν τα μοχλευόμενα επενδυτικά κεφάλαια είναι πιο ευαίσθητα στις αλλαγές, στις αλλαγές των τιμών, στις πιέσεις, οπότε μπορεί να οδηγηθούμε σε απομόχλευση με πώληση παγιών στοιχείων για να έχουμε ρευστότητα. Αυτό αν γίνει απότομα θα υπάρχει κίνδυνος ε, στη ρευστότητα ο οποίος μπορεί να επεκταθεί και σε άλλες αγορές. Γι' αυτό πρέπει να βρούμε τους συστημικούς κινδύνους που τίθενται ε, όποτε τα επενδυτικά κεφάλαια εκτίθενται σε αυτούς τους κινδύνους. Αυτή είναι μία από τις δικές μας δουλειές. Ελπίζω σύντομα να έχω να σας πω περισσότερα. Αυτό μαζί με το γεγονός ότι έχουμε μία κυκλική δραστηριότητα στον ε, τομέα τον οικονομικό ε, μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη χρήση των παραγόγων και τις συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων. Οι συναλλαγές σε παράγωγα, ο πιστοτικός κίνδυνος αντιστημβαλόμενου μειώνονται, ενώ οι πρόσθετες εξασφαλίσεις παίζουν περισσότερο, μεγαλύτερο ρόλο στη συναλλαγή χρηματοδότησης τίτλων. Τα κουρέματα λοιπόν μπορεί να προστατεύουν τους αντισυμβαλόμενους και τα περιθώρια βοηθούν στην απορρόφηση των απολειών, βοηθώντας επίσης και τη διαχείριση του χρηματοπιστωτικού κινδύνου. Για, επίσης μειώνουν την συσσόρευση της ηρωή μόχλευσης. Για παράδειγμα, ε, τα κουρέματα ορίζουν και το ποσό της χρηματοδότησης που μπορεί να πάρει κανείς από μια εξασφάλιση. Τα περιθώρια επίσης μπορεί να δρουν με βάση τον κύκλο της οικονομίας σε χαμηλότερα επίπεδα και σε ευνοϊκούς καιρούς επιτρέπουν την συσσόρευση μόχλευσης. Όταν αυξάνονται κατά την ύφεση μπορεί να οδηγήσουν σε αρνητικά σπιράλ. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν το Συμβούλιο χρησιμοποιεί μακροπροληπτικά εργαλεία τα οποία στοχεύουν στα περιθώρια και στο κούρεμα επίσης ε, προσπαθούμε να βρούμε ποιες είναι οι πρακτικές προκλήσεις κατά την εφαρμογή των εργαλείων. Το, banking, το Shadow Banking Monitor ε, βρίσκει ποια είναι η διασυνδεσιμότητα και ο κίνδυνος ε, μετάδοσης ε, σε διάφορα τμήματα του χρηματοπιστωτικού τομέα και εντός του συστήματος μη τραπεζικών συναλλαγών. Αυτή η διασυνδεσιμότητα είναι ένα γενές στοιχείο ενός ολοκληρωμένου χρηματοπιστωτικού συστήματος και αντικατοπτρίζει τις ροές ε, χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης. Έχει διάφορες μορφές και γι' αυτό πρέπει να παρακολουθείτε για να αποφύγουμε την μετάδοση σε περίοδους ε, μεγάλης, ε, μεγάλου στρες. Έτσι λοιπόν ο κανονισμός ΕΜΙΡ για τις υποδομές των ευρωπαϊκών αγορών μας έδωσε πρόσβαση σε ολοκληρωμένα στοιχεία για τις συναλλαγές σε παράγωγα. έχουμε μια ευρωπαϊκή εικόνα και γι' αυτό ε, βασιζόμαστε στα στοιχεία αυτά έτσι ώστε να βρούμε ποιες, ποιες είναι οι σχέσεις μεταξύ μη τραπεζικών συναλλαγών και αγορών παραγόγων. Υπάρχουν τρεις μεγάλες αγορές, ε, π.χ. Ε, επιτόκια, συνάλλαγμα και παράγωγα πιστοτικά που αντιστοιχούν με 7, 19 και 10%. Επίσης, η έκθεση εξετάζει το τοπίο των αντισυμμαλόμενων στον τομέα αυτών. Δείχνει επίσης η έκθεση ότι το 60% της έκθεσης των Ευρωπαϊκών Τραπεζών σε μη τραπεζικές ε, οντότητες ε, είναι σε οντότητες που δεν έχουν την έδρα τους ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι αυτό που είπαμε πριν για τα CCP και το Euroclearing. Συγκεκριμένα η ανάλυση δείχνει το στενό δεσμό μεταξύ Ευρωπαϊκών Τραπεζών και οντοτήτων που βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες και ε, κάνουν, εκτελούν συναλλαγές ε, μη τραπεζικές. Αυτά τα ευρήματα λοιπόν μας καταδεικνύουν την ανάγκη διεθνούς συνεργασίας και παρακολούθησης. Το πλαίσιο λοιπόν έχει εποφεληθεί από τις πρόσφατες μεταρρυθμίσεις ε, και τις εξελίξεις στον τομέα των δεδομένων. Αλλά παραμένουν οι προκλήσεις και χρειάζονται περισσότερες προσπάθειες για να κλείσουμε τα υφιστάμενα κενά που αφορούν ε, στον ε, διασυνοριακό και διατομεακό τομέα. Να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη άποψη για τη μη τραπεζική πιστοτική δραστηριότητα επιπλέον, δηλαδή ε, θα, πρέπει, θα μπορούσαμε να υποφεληθούμε και από δεδομένα τα οποία διατίθεται και σε επίπεδο ε, ενοποιημένο ή μη ενοποιημένο. Νομίζω ότι σας έδωσα μια γενική άποψη για αυτή την έκθεση. Να καταλήξω τώρα με κάποιες παρατηρήσεις γενικά για την μακροπροληπτική πολιτική έχει γίνει μεγάλη πρόοδος στην ανάλυση του μη τραπεζικού τομέα. Να σας δώσω ένα ακόμα παράδειγμα. Η ΟΠΑ έκανε ε, τα πρώτα στρες για τις επαγγελματικές συντάξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2015 και πρόσφατα ξεκίνησε το δεύτερο τεστ, στο οποίο το Συμβούλιο μας συνεισέφερε ε, ε προετοιμάζοντας ένα ε, σενάριο μη ευνοϊκό. Παρόλα αυτά, ε, είμαστε ακόμα σε πρώιμο στάδιο, χρειαζόμαστε κάποια εργαλεία, κάποια μέσα, ε, πέρα από αυτά που έχουμε που είναι για συγκεκριμένο σκοπό, για να έχουμε μια πλήρη εργαλειοθήκη. Έχω αναφέρει κάποια εργαλεία από αυτά. Ήδη τα περιθώρια, οι απαιτήσει περιθωρίων και κουρέματος. Επιπλέον, ε, η μορφή των καθεστώτων εξυγίανσης ε, για τους κεντρικούς αντισυμβαλόμενους ε, και τις ασφαλιστικές εταιρείες θα πρέπει να έχει ένα προφίλ μακροπροληπτικό. Το Συμβούλιο μας έχει θέσει αυτά τα θέματα ε, στην απάντησή του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν αυτή ξεκίνησε τη σχετική διαβούλευση. Τώρα θα σας μιλήσω για το γεγονός ότι τα εθνικά θεσμικά πλαίσια για τη μακροπροληπτική πολιτική έχουν μεγάλη σημασία για να είναι αποτελεσματική αυτή η πολιτική. Σε δύο κράτη-μέλη έχουμε μια νομοθετική διαδικασία η οποία συνεχίζει και έχει να κάνει με την μακροπροληπτική αρχή έχουν ήδη χρησιμοποιήσει τα ε, διαθέσιμα εργαλεία του το 2016 οι αρχές, ε, σύμφωνα με την ε, οδηγία CRD4 και CRR. Πρόσφατα το Συμβούλιο μας έκανε, δημοσίευσε μια γενική επισκόπηση των μακροπροληπτικών πολιτικών, όπου αναφέρονται όλα αυτά τα μέτρα που υιοθετήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2016. Ευχαριστώ πολύ. Λόγω περιορισμένου χρόνου ε, θα πρέπει να ομαδοποιήσουμε τις ερωτήσεις και η κάθε ερώτηση να είναι το πολύ 1,5 λεπτό. Πρώτη ερώτηση ο κύριος Κίρτσος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήθελα να ρωτήσω τον πρόεδρο Ντράγκη την άποψή του, για την άποψή του σχετικά με τον τι κίνδυνο παρουσιάζει ο τραπεζικός, το τραπεζικό ελληνικό σύστημα. Είχαμε κάποιε εξελίξει θετικέ, αρνητικέ, που πρέπει όμω να αξιολογηθούν. Παραδείγματο χάρη, ε, τα κόκκινα δάνεια παραμένουν σε πολύ υψηλό επίπεδο. Είχαμε και μια τρομοκρατική επίθεση κατά του κ. Παπαδήμου, του πρώην Έλληνα Πρωθυπουργού, πρώην κυβερνήτη της Τράπεζας της Ελλάδας και αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ίσως να στέλνετε ένα μήνυμα έτσι από τους τρομοκράτες κατά της αναδιάθρωσης των τραπεζών και της ε, διαχείρισης ε, αυτών των δανείων. Από την άλλη κάποιες τράπεζες είναι πολύ κοντά στο να έχουν κέρδη και έχει αυξηθεί σημαντικά ε, και η αξία των μετοχών τους τους τελευταίους μήνες. Εσείς πιστεύετε ότι ο συστημικός κίνδυνος θα ελεγχθεί και το τραπεζικό σύστημα ε, θα μπορέσει να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας στο προσεχές μέλλον ή θα επαναλάβουμε τα προβλήματα του παρελθόντος που οδήγησαν στην ανακεφαλοποίηση του τραπεζικού κλάδου. Ευχαριστώ. Ναι, σου μπερές τώρα, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μόλις ε, δημοσίευσε τις προτάσεις της ε, για την ενιαία αγορά κεφαλαίων και έχει προσθέσει και μία διάσταση έτσι ανησυχητική ό,τι αφορά τη μακροοικονομική σταθερότητα. Εσείς ε, θεωρείτε ότι έχετε όλα τα εργαλεία στη διάθεσή για να αντιμετωπίσετε ε, κάποιες εξελίξεις, κάποιες κινήσεις στην αγορά μη επιθυμητές, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την τιτλοποίηση, μπορείτε να παρέμβετε εφόσον έχουμε εξελίξεις με φούσκες τη μία ή την άλλη χώρα και όπως προτείνουμε και στη διαπραγμάτευση που είναι εξελίξη η προσαρμογή του ποσοστού ε, παρακράτησης ανάλογα με την ποιότητα του δανειστή πιστεύετε ε, ότι είναι ενδιαφέροντα εργαλεία, σημαντικά εργαλεία για να μπορείτε να παρέμβετε για να επιτευχθεί ο στόχος της σταθερότητας. Ο Νότης Μαριάς έχει το λόγο, παρακαλώ. Κύριε με το τρίτο δανειακό πακέτο είχε προβλεφθεί ποσό 25 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Όμως χρησιμοποιήθηκαν μόνο 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ για την ανακεφαλαιοποίηση. Έχουν περισσέψει λοιπόν αυτή τη στιγμή 19,5 δισεκατομμύρια ευρώ από το τρίτο δανειακό πακέτο. Ταυτόχρονα υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα με τα κόκκινα δάνεια, τα NPLs. Με αποτέλεσμα πολλοί Έλληνες να κινδυνεύουν πλέον να χάσουν τα σπίτια τους μια και τα distress funds πλέον ε, έχουν πάρει, έχουν αγοράσει πολλά δάνεια και μάλιστα τα έχουν αγοράσει στο 10% της αξίας τους. Συμφωνείτε να δημιουργηθεί ένα δημόσιο ταμείο για κόκκινα δάνεια με 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ από, τα υπόλοιπα των 19,5 που είχαν προβλεφτεί για την ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών και αυτό το δημόσιο ταμείο για τα κόκκινα δάνεια να στηρίξει τους δανειολήπτες να μπορέσουν να πληρώσουν το δάνειό τους για να μην αρπάξουν τα κοράκια τα σπίτια τους και μάλιστα να εφαρμόσουμε στην Ελλάδα και το μοντέλο της Κύπρου δηλαδή να έχουν δικαίωμα οι δανειολήπτες αυτοί οι ίδιοι σαν πρώτη προσφορά να έρθουν να πληρώσουν το δάνειό τους στην τιμή προσφοράς που θα, τους κάνουν, που θα τα distress funds στις τράπεζες. Ευχαριστώ. Cora van Leeuwenhuizen. Cora van Leeuwenhuizen. Chair, um, well, welcome to you again, Mr. Ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε εκ νέου, κύριε Ντράγκη. Ένας από του μεγαλύτερου κινδύνους που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή έχει να κάνει με τις κυβερνοεπιθέσεις. Είχαμε την ε, επίθεση του ransomware η οποία ήταν σχετικά ε, ανώδυνη, αλλά το όλο σύστημα τραπεζικό βασίζεται στην σύνδεση, στα δεδομένα, στο διαδίκτυο. Εσείς πιστεύετε ότι στη δική σας οργάνωση, αλλά και στις εθνικές αρμόδιες αρχές δίνεται επακής προτεραιότητα στην κυβερνοασφάλεια. Εσείς πιστεύετε ότι θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προτεραιότητα στα stress test των τραπεζών, διότι εξαρτώμεθα όλο και περισσότερο από την ψηφιοποίηση. Ένα δεύτερο ερώτημα τώρα που έχει να κάνει με, το CCP, με CCP και το clearing, με το παρόν πολιτικό κλίμα. Όταν μιλάμε για μετεγκατάσταση ε, του clearing των ευρώ, ε, δεν θα μπορούσε ε, οι Ηνωμένε Πολιτείε να ζητούν να υπάρχει καθάριση δολαρίων μόνο στι Ηνωμένε Πολιτείε ω αντίπεινα. Και είχα και ένα άλλο ερώτημα, αλλά δεν ξέρω, κοιτάζω και τον πρόεδρο, θα το ρωτήσω, θα το ρωτήσω άλλη φορά. Μάλιστα, πολύ ωραία. Και ο κύριος Παπαδημούλης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Ντράγκη, θα σας ρωτήσω για τη χώρα μου, την Ελλάδα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανήκει στο κουαρτέτο των δανειστών. Και όλες οι επίσημες δηλώσεις και οι δικές σας λένε πως διαφαίνεται μια ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας για τα επόμενα χρόνια και ότι χρειάζεται μεγαλύτερη εμπιστοσύνη και καθαρός οδικός ορίζοντας έτσι ώστε να μπορέσει μετά τον Αύγουστο του 2018 και η χώρα μου η Ελλάδα να μπορεί να δανείζεται από τις αγορές με λογικά επιτόκια χωρίς μνημόνια και δάνεια. Το ερώτημά μου είναι από τη στιγμή που εκφράσατε τη λύπη σας γιατί δεν ολοκληρώθηκε αυτή η συμφωνία στο Eurogroup της 22ης Μαΐου. Τι περιμένει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και εσείς προσωπικά από το επόμενο Eurogroup στις 15 Ιουνίου προκειμένου να προχωρήσει, να αποσαφινιστεί αυτός ο οδικός χάρτης όπως τον έχετε υποσχεθεί για να μπορέσετε κι εσείς να κάνετε τη δική σας αξιολόγηση και να εντάξετε στο άμεσο μέλλον και την Ελλάδα στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. Ως πότε η ελληνική οικονομία και ο ελληνικός λαός θα πληρώνουν την ανελαστικότητα και την αναβλητικότητα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της κυβέρνησης του Βερολίνου. Η Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το Ευρωκοινοβούλιο, το Eurogroup, η ελληνική κυβέρνηση θέλουν συμφωνία και καθαρό οδικό χάρτη. Πότε επιτέλους θα σταματήσει αυτή η διαρκής αναβολή. Um, Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω πρώτα τα ερωτήματα για την Ελλάδα. Παρόλο που η Ελλάδα δεν συζητήθηκε ξεκάθαρα σε καμία από τις συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικών Κινδύνων πρόσφατα και τον τραπεζικό τομέα Πραγματικά έχει γίνει εξαιρετική πρόοδος, αξιοπρόσεκτη πρόοδος, ειδικά αν δούμε την κεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών σήμερα. Δεν έχω ακριβώς το νούμερο, όμως είναι πολλαπλάσια από ό,τι ήταν πριν. Εν τούτης, ε, έχουμε πολύ μεγάλο ποσοστό κόκκινων δανείων. Τέθηκε αυτό το ερώτημα και αυτό εν μέρη οφείλεται στην κρίση αλλά και σε προϋπάρχουσες αδυναμίες του πιστοτικού τομέα. Ε, υπάρχουν πολλές δράσεις που προβλέπονται στο τρέχον πρόγραμμα και είναι απαραίτητες για να είναι επιτυχημένη η κατάληξη της ε, αξιολόγησης. Αυτές οι δράσεις ε, αφορούν σε πράγματα που πρέπει να κάνει η κυβέρνηση, οι τράπεζες, ε, να υπάρξει ένα εξοδικαστικό πλαίσιο για την ε, ε, διάθεση των κόκκινων δανείων. Οι χώρες παρεπιπτόντος που δεν έχουν ένα πλαίσιο για την εύκολη διάθεση των κόκκινων δανείων ή έχουν μια δικαστική διαδικασία η οποία είναι βραδία και αναποτελεσματική ή μια νομοθετική διαδικασία ε, που επιβραδύνει όλα αυτά είναι αυτές που έχουν και τα υψηλότερα επίπεδα κόκκινων δανείων. Σε πολλές χώρες το πρόβλημα αυτό παραμένει εδώ και χρόνια, δηλαδή δημιουργήθηκε ένα απόθεμα τέτοιων δανείων από το παρελθόν και τώρα αποτελούν πρόσκομα στις δραστηριότητες των τραπεζών και υπάρχουν και χώρες οι οποίες λύνουν το πρόβλημα των καινούριων κόκκινων δανείων και όχι τα παλιά. Αυτό βέβαια δεν είναι η περίπτωση της Ελλάδος. Πρόκειται λοιπόν για ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει το τρέχον πρόγραμμα με την τρέχουσα αξιολόγηση και αν ε, ε, λάβουν χώρα οι δράσεις που προβλέπονται σε αυτό θα επιληθεί εγκαίρως το πρόβλημα. Αναφέρεται το Λουκά Παπαδήμο παρεπιπτόντος υπήρξε εξαιρετικός αντιπρόεδρος της ΕΚΤ, εξαιρετικός πρωθυπουργός και είναι πολύ πολύ καλός μου φίλος. Και θα ήθελα να εκφράσω την αλληλεγγύη μου, τα τρυφερά μου συναισθήματα, προσωπικά εγώ, αλλά και εκ μέρους ε, του προσωπικού της ΕΚΤ, ε, του Εκτελεστικού Συμβουλίου και του Διοικητικού Συμβουλίου. Συνεχίζοντας για την Ελλάδα, να πω ότι περιμένω από το επόμενο Ευρω... Eurogroup. Η απάντηση, μάλλον η συμφωνία σχετικά με το χρέος, ποια είναι τα μέτρα που θα καταστήσουν το χρέος βιώσιμο για την Ελλάδα, είναι ένα θέμα που έχει συζητηθεί από τη μία μεταξύ των κρατών μέλων και από το δούνου του από την άλλη. Φτάσαμε λοιπόν σε ένα σημείο που τα δύο μέρη θα πρέπει να βρουν ένα κοινό σημείο, μια συμφωνία. Αυτό χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή. Να προσθέσω επίσης ότι η ποσοτική χαλάρωση για την Ελλάδα δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Πρέπει να κάνουμε και εμείς τη δική μας ανεξάρτητη αξιολόγηση και βάση ε, αντίξων σεναρίων βιωσιμότητας. Πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη διάφορα στοιχεία. Να ξεκαθαρίσω όμως ότι η αξιολόγηση βιωσιμότητας του χρέους που κάνει η Κομισιόν, το ΔΝΤ, η ΕΚΤ, δεν σημαίνει ότι και η επόμενη ε, αξιολόγηση θα είναι ίδια. Τώρα, για τα μακροοικονομικά, χρηματοοικονομικά μέσα που είναι διαθέσιμα για την ε, ε, ενιαία αγορά ε, κεφαλαίων στην Ευρώπη έχουμε πει ότι είμαστε υπέρ της διαφοροποίησης των πηγών χρηματοδότησης. Όμως πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι αυτοί που χαράσουν την πολιτική πρέπει να έχουν τα εργαλεία για να μπορέσουν να προλάβουν και να μετριάσουν το συστημικό κίνδυνο που θα που ενδεχομένως να ανακύψει σε αυτήν την ένωση κυρίως ε, στον τομέα της μη τραπεζικής πιστοτικής δραστηριότητας, το shadow banking. Ε, βλέπουμε πόσο μεγάλη ανάπτυξη έχει αυτός ο τομέας και συζητήσαμε πριν το fintech, δηλαδή την οικονομική τεχνολογία ε, που αποτελεί κομμάτι αυτού του τομέα. Πρέπει λοιπόν να υπάρχουν εργαλεία μακροπροληπτικής εποπτείας και γι' αυτό το θέμα είδαμε ότι υπάρχει μια ε, αναθεώρηση του κανονισμού για το ESA και ενίσχυση του ΕΣΜΑ. Επομένως, ε, ε, θα συνεχίσουμε να έχουμε τα μάτια μας σε αυτό το θέμα. Υπάρχουν βέβαια διάφορα μέτρα που θα μετριάσουν την ε, ικανότητα σύναψης νέου χρέους οτιδήποτε δηλαδή έχει να κάνει με την πλευρά της ζήτησης για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα, ε, τα μακροπροληπτικά στον τομέα μη τραπεζικής πιστοτικής δραστηριότητας. Το ερώτημα για τις κυβερνοεπιθέσεις. Ναι, όντως ε, πρέπει να δώσουμε μεγάλη προτεραιότητα στην κυβερνοασφάλεια. Αυτή τη στιγμή έχουμε συνειδητοποιήσει πλήρως ότι αυτό ενδεχομένως να είναι το πιο σημαντικό ή μάλλον είναι το πιο σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι αρχές μας. Στην τελευταία συνάντηση G7 οι Υπουργοί Οικονομικών ακριβώς αυτό συζήτησαν. Παρεμπιπτόντως σε όλα τα διεθνή βήματα συζητιέται αυτό το ζήτημα, φυσικά στην ΕΚΤ και φυσικά στις εθνικές αρμόδιες αρχές. Τώρα για τα stress test ε, στις τράπεζες όσον αφορά στην κυβερνοασφάλεια. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα, το έκανε η Τράπεζα της Αγγλίας και χαιρετίζουμε τυχόν πρωτευουλίες από τις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες και Εποπτικές Αρχές στην Ευρωζώνη. Εμείς κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση και θεωρούμε ότι είναι κάτι που ε, εμπίπτει στον τομέα των stress tests. Τώρα η πολιτική μεταγκατάστασης. Όπως είπα και πριν, είναι πολύ δύσκολο να πούμε ποια θα είναι η τελική συμφωνία που θα βρουν τα διάφορα μέρη, διότι εμείς δεν είμαστε μέρος σε αυτή τη την συμφωνία. Μπορούμε όμως να δώσουμε συμβουλές. Όποια όμως και αν είναι η συμφωνία, το σημαντικό για μας είναι να έχουμε σημαντική εξουσία εποπτείας, ελέγχου των δραστηριοτήτων ε, ε, clearing ε, του ευρώ και των δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή, στον Ευρωζώνη. Δεν απαντήσατε την ερώτηση για τα κόκκινα δάνεια στην Ελλάδα. το ποσό που απομένει από την αναδιάρθρωση των τραπεζών. Σας είπα ότι η Ελλάδα δεν συζητήθηκε, δεν ξέρω. Πραγματικά δεν έχω ιδέα τι θα κάνουμε με αυτό το ποσό. Αυτή είναι η απάντηση που έχω να σας δώσω. Εδώ ε, η ακρόαση είναι για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικών Κινδύνων. Το θυμίζω. Φίλιπ Λάμπερτς. Δεν τον βλέπω. Πάρε Κάπελ. Ευχαριστώ, Κύριε Διοικητά, αναφερθήκατε στην επιτήρηση του τομέα των σκιωδών τραπεζικών δραστηριοτήτων και το σημαντικό κομμάτι του οικονομικού κλάδου που καταλαμβάνουν αυτές. Στην έκθεση λοιπόν αυτή, έκθεση υποπτία σημειώνεται ένα πρόβλημα σε σχέση με την επικαιρότητα των στοιχείων Ιδιαίτερο για τις σκιώδεις τραπεζικές δραστηριότητες από την Κίνα, γιατί είναι το 2010. Έχετε λοιπόν πιο πρόσφατα στοιχεία, έχετε συνεργασία ενδεχομένω με τις κινέζικες αρχές για να έχετε τα στοιχεία που απαιτούνται για το monitoring αυτό. Έχετε ενδεχομένω στοιχεία από τρίτες πηγές για να συμπληρώσετε τη, τα δεδομένα σας. Και επίσης άλλη μια ερώτηση που έχει να κάνει με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ε, εποπτεία της μακροληπτικής εποπτείας που μας αναφέρατε και εσείς ότι δύο χώρες δεν έχουν τέτοιου είδους αρχές. Η μία είναι η Ιταλία πιστεύω. Ε, έχουν βγει βέβαια κάποια εκτελεστικά διατάγματα και θέλω να ρωτήσω αν έχετε ορίσει ένα ε, χρονοδιάγραμμα για τα εκτελεστικά διατάγματα, ειδικά για την Ιταλία, για την εισαγωγή αυτής της αρχής και δεύτερον τι προτεραιότητες έχετε ορίσει για την μακροληπτική εποπτεία, ειδικά για την Ιταλία πάλι. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος. Βάλλη. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ντράγκη, έχω για σας μια ερώτηση. που αφορά το Συμβούλιο, αλλά βεβαίως και την έκτη γενικότερα. Σε μια χρονική στιγμή όπου βρισκόμαστε σε μια περίοδο πιθανολογούμενης εξόδου από το QE, και αύξηση των επιτοκίων, ε, τίθεται πιο πιεστικά το ζήτημα του κρατικού χρέους ορισμένων κρατών και δι της Ιταλίας. Βεβαίως εδώ έχουμε μηχανισμούς οι οποίοι δεν προσφέρουν δεν στηρίζονται σε μια βάση αλληλεγγύης, αλλά περισσότερο σε μια διαδικασία με την οποία ε, ο, τα ομόλογα από ορισμένε χώρες θα μπορούσαν να κατανέμονται ανάλογα με διαφορετικά προφίλ κινδύνου. Ένα νέο εργαλείο λοιπόν το οποίο όμω θα εντείνει φοβούμαστε τον κατακαιρματισμό και τις διαφορές μεταξύ των κεντρικών και των περιφερειακών χωρών και ιδιαίτερω για τις χώρες τη της θα εντείνει την παρουσία και άρα του κινδύνου σε σχέση με τι ε, ε, κεφαλαιακές δυνατότητες και βάσει των τραπεζών. Ε, υπάρχει δυνατότητα για μεγαλύτερο επιμερισμό του κινδύνου, γιατί δεν βλέπω αυτή τη στιγμή δυνατότητα να μείνει βιώσιμο το χρέος σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Και ξέρω ότι είστε ε, ακρεφνής φιλοευρωπαίος. Θέλω λοιπόν τη γνώμη σας γι' αυτό. Κύριο Τόμας Μαν. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριε Ντράκη, στην ομιλία σας Ε, θα ήθελα να σταθώ λίγο στο τελευταίο σημείο που έχει να κάνει με την ε, πολιτική των ακινήτων και τα ακίνητα. Είδαμε λοιπόν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από ό,τι μας είπε ο ε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου. Μας είπε ότι δεν βλέπει κίνδυνο φούσκας στην αγορά των ακινήτων. Ωστόσο, είναι πολύ σημαντική η κίνδυνη να ενισχυθούν υπέρ το δέον οι τιμές των ακινήτων. Είναι πολλοί αυτοί που παίρνουν δάνεια τώρα γιατί έχουν χαμηλά επιτόκια. Και ο Ανδρέας Δόντρε που έκανε μια ομιλία πρόσφατα στην ε, Βουλή ναι, είπε ότι αυτή τη στιγμή είναι στο κίτρινο το φανάρι, στο πορτοκαλί το φανάρι ε, για την πορεία της αγοράς των ακινήτων. Πώς μπορεί λοιπόν το Συμβούλιο να αξιολογήσει την κατάσταση αυτή και δεν αναφέρομαι μόνο στη Γερμανία αλλά γενικότερα στην Ευρώπη στην αγορά των ακινήτων. Κύριε κύριος Φερνάντες, τελευταία ερώτηση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κύριε Ντράγκη που είστε εδώ μαζί μας. Δύο ερωτήσεις πολύ σύντομα. Ε, η πρώτη έχει να κάνει με αυτήν που έθεσε και η κυρία Μπερές προηγουμένως ό,τι αφορά τις για την τυπλοποίηση STS ε, διαπραγματευόμαστε με το Συμβούλιο αυτή τη στιγμή ένα κείμενο το οποίο δίνει τη δυνατότητα να υπάρχει μία ε, εποπτεία μακροπρόθεσμη της συγκεκριμένη αγοράς το ESRB θα πρέπει να μπορεί να ε, εξετάζει το, το risk retention ε, πιστεύετε ότι θα μπορείτε να κάνετε κάτι τέτοιο αυτός ο οργανισμός ο δικός σας δηλαδή αναφερθήκατε επίσης νωρίτερα ε, στο θέμα των κόκκινων δανείων στην Ελλάδα ε, υπάρχει μια ομάδα εργασίας που εξετάζει την δυνατότητα να δοθεί μια ευρωπαϊκή απάντηση για τα κόκκινα δάνεια πώς πάνε οι εργασίες της ομάδας Uh, θα απαντήσω στις απαντήσεις Ελπίζω να θα τηρήσω και τη σειρά με την οποία τυπώθηκαν. Για, για την Κίνα. Η κυβέρνηση της Κίνας δεν δίνει πολύ λεπτόμερα ε, στοιχεία, ούτω ή άλλως δεν μας ενδιαφέρουν. Ε, ευρωπαϊκά στοιχεία ε, χρειαζόμαστε εμείς. Για την Ιταλία έχει περάσει σχετική νομοθεσία η Ιταλική κυβέρνηση τώρα στη διαδικασία της ε, θέσης εφαρμογή του σχετικού νόμου. Το Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου για τη SB έχει μια task force ή καλύτερα είναι μια δομή που ξεκινάει τη συζήτηση αυτή. Task force υπό τον διοικητή Φίλιπ Λέιν της ε, Κεντρικής Τραπεζής της Ιρλανδίας Και για να το πω περιφραστά, το ΙΣΠ είναι μία πρόταση με βάση την οποία θα γίνεται μια ε, ομαδοποίηση και μια σύνθλιψη των ε, ομολόγων, χωρίς αυτό όμως να σημαίνει ε, επιμερισμό του κινδύνου. Δηλαδή δεν αντικαθιστά με κάποιο τρόπο τα ευρωομόλογα. Είναι κάτι το διαφορετικό, απλούστατα. Και έτσι η ΕΚΤ, όχι το Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου, η ΕΚΤ με το Διοικητικό Συμβούλιο καταγράφει αυτή την εξέλιξη και θα έλεγα ότι είναι πολύ νωρί. Δεν μπορούμε δηλαδή να καταλήξουμε προ τη μία την άλλη κατεύθυνση σε θέσει για την ιδέα αυτή. Προ το τέλος του τρέχοντο έτου, μάλλον προ τον Νοέμβριο θα δούμε μια τελική έκθεση για τις κατοικίε και τα ακίνητα. Τα ακίνητα λοιπόν για κατοικία παρουσιάζουν αύξηση τιμών, ιδιαίτερα στις μεγάλες, στα μεγάλα αστικά κέντρα της Γερμανίας, αλλά και στις κάτω χώρες, στην Αυστρία και άλλες χώρες. Και το Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου έχει εκδώσει προειδοποίησεις προς την κατεύθυνση αυτή, τις οποίες μάλιστα συζητήσαμε και στη τελευταία μας ακρόαση. Τώρα να κοιτάξουμε τις ε, Δηλαδή, εάν περάσουμε ε, πέραν των αστικών, μεγάλων αστικών κέντρων και κοιτάξουμε τη γενικότερη εικόνα σε μια χώρα, εάν εν γέννη δηλαδή ε, παρουσιάζει αυξητικέ τάσει ο κλάδος των ακινήτων στις ορισμένες χώρες, ο μέσος όρος μένει λίγο πολύ στου στους μέσου μέσους όρους. Δεν βλέπουμε δηλαδή μια υπερβολική αύξηση τιμών συστημικού χαρακτήρα. Αύξηση τιμών βλέπουμε σε ε, συγκεκριμένες τοπικές αγορές, αλλά όχι σε συστημική βάση. Και επιτρέψτε μου επίση να συμπληρώσω ότι ενώ αυξάνονται οι τιμέ των ακινήτων, δεν βλέπουμε να αυξάνεται ο πιστοτικό όγκο με του ίδιου ρυθμού. Ούτε καν σε συγκρίσιμου ρυθμού σε σχέση με αυτό που είχαμε πριν από την κρίση. Δηλαδή, τα δάνεια ενυπόθηκα δάνεια, η κτηματική πίστη δεν ε, βλέπουμε να έχει σημαντική ε, αύξηση. Εν πάση περιπτώσει βλέπουμε σε ορισμένες χώρες και σε μία που έχω υπόψη το φαινόμενο πολλοί ιδιοκτήτες ακινήτων να βρίσκονται σε κατάσταση αρνητικού ενεργητικού με την έννοια ότι η τιμή, η αξία των σπιτιών τους είναι υψηλότερη από αυτή του χρέους τους. Και βέβαια αυτό θα πρέπει να αντιστραφεί. Για τη διασφάλιση. Τιτλοποίηση. Βεβαίως ε, θα πρέπει να κάνουμε μια επισκόπηση ως ε, Συμβούλιο των Μακροληπτικών ε, Συνθήκων. Και τελευταίο σημείο βεβαίως παρακολουθούμε τις συζητήσεις που διεξάγονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχέση με την τιτλοποίηση και συμφωνούμε σε μεγάλο βαθμό απλώς ιδιαίτερο μέλημα έχουμε την αύξηση των ε, λόγων διακράτησης χρέους, γιατί θέλουμε να έχουμε τη δυνατότητα να το ξαναρίξουμε όλο αυτό στην πραγματική οικονομία και πιστεύουμε ότι τα χαρακτηριστικά των ε, εργαλείων που είναι υποσυζήτηση ε, είναι αρκετά ασφαλή. Ένας υπερβολικά υψηλός κίνδυνος διακράτησης θα μπορούσε να εμποδίσει την ε, διασπορά και την επιτυχία των εργαλείων αυτών. Για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Βεβαίως, το είπαμε, και νωρίτερα οι δράσεις που προβλέπονται στο πρόγραμμα της Ελλάδας αφορούν δράσεις από πλευράς των, των τραπεζών για τη διαχείριση του κινδύνου και την ανάκτηση του χρέους. Πρέπει από εκεί και πέρα η διακυβέρνηση να εξασφαλίσει ένα περιβάλλον το οποίο να ε, διευκολύνει την διάθεση των δανείων με αλλαγές στις δικαστικές διαδικασίες, στους εξαδικοστικούς συμβιβασμούς και μια σειρά ακόμη δράσεων που μας οδηγούν στο συμπερασμό τη δημιουργία μία τέτοιας εταιρείας διαχείρισης ε, ενεργετικού μπορεί να είναι μία λύση, αλλά δεν μπορεί να είναι η μία και μοναδική λύση σε εθνικό επίπεδο, όπως άλλωστε δεν μπορεί να είναι η μία και μοναδική λύση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Με μεγάλο ενδιαφέρον λοιπόν παρακολουθούμε τις εξελίξεις αυτές, αλλά δεν πιστεύουμε ότι κάτι τέτοιο θα αρκέσει όλες οι άλλες δράσεις. Επόδυνες πολλές φορές είναι οι απαραίτητες δράσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Κλείνουμε εδώ και αυτή τη δεύτερη ακρόαση. Πάντα πολύ χρήσιμη και ενδιαφέρουσα. Ευχαριστώ τον διοικητή, τον κύριο Ντράγκη για την παρουσία του, γιατί είναι όπως πάντα πολύ θετική και ε, επικοδομητική συζήτηση και το συνεχή διάλογο.